So, και ένα. Αρχίζουμε. Start. Uh, we will uh, switch to point 12. Θα περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η παρουσίαση μελέτης για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit. Έχουμε εδώ τον καθηγητή Eckhout μαζί μας, ο οποίος ε, έχει συντάξει και τη μελέτη αυτή και ο οποίος θα μας την παρουσιάσει σε 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την μελέτη που συντάξαμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε και να τη δημοσιεύσουμε για το Κοινοβούλιο και να σας την παρουσιάσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στην παρουσία μου, να μην σας παρουσιάσω όλα τα σημεία στα οποία αναφέρεται η έκθεση αυτή, η μελέτη αυτή αλλά θα βασιστώ στα κύρια στοιχεία. Εννοείται ότι πρόκειται για κινούμενο στόχο, έτσι, το Brexit. Μπορεί να μην είναι αυτό καθ' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι όλα αλλάζουν από πλευράς, αν μη τι άλλο, του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια μελέτη που ολοκλήρωσα τον Φεβρουάριο και σε ένα βαθμό φαίνεται να έχει ήδη ξεπεραστεί για κάποια ζητήματα όσον αφορά τους διακανονισμούς για μετά το Brexit. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δούμε ποια είναι τα πρότυπα που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί σχολιαστές εξέτασαν τα διάφορα εμπορικά μοντέλα για μετά το Brexit, προσπαθώντας να αποφασίσουν πού θα καταλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένων των σχέσεων που έχει, δεδομένων ε, των δεσμών που έχει με διάφορες ε, χώρες, ε, το νορβηγικό μοντέλο, το τουρκικό, το τουρκικο το ολβετικο κλπ. Πιστεύω όμως ότι εκτός από αυτά τα μοντέλα υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο και αυτή ακριβώς είναι η δυσκολία, δηλαδή η ολοκλήρωση της αγοράς. Ποια θα είναι η σχέση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την Ελβετία, με την Ουκρανία και από την άλλη έχουμε και την απελευθέρωση του εμπορίου. Είναι και αυτό ένα άλλο πρότυπο το οποίο έχει και αυτό αναπτυχθεί και εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μία και στην άλλη περίπτωση και συζητιούνται όλα. Εγώ προσπάθησα να επικεντρωθώ περισσότερο σε αυτά που εγώ γνωρίζω καλύτερα, δηλαδή τις νομικές και θεσμικές διαφορές ανάμεσα στην ολοκλήρωση της αγοράς και την απελευθέρωση του εμπορίου. Τα τελευταία 20 χρόνια, αν δούμε πώς εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής εμπορική πολιτική, οι διεθνείς εμπορικές ε, σχέσεις, διαπιστώνουμε ότι το χάσμα έχει μεγαλώσει ανάμεσα σε μια ολοκληρωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απελευθέρωση του εμπορίου. Η μελέτη μου δεν σχολιάζει καθόλου τις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά τα οικονομικά μοντέλα δύσκολα μπορούν να λάβουν υπόψη τους τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο μοντέλα. Και θα ανησυχούσα πάρα πολύ για αυτό το επίπεδο αβεβαιότητας που δημιουργείται για τους επενδυτές αν εγκατέλειπε το μοντέλο της ολοκληρωμένης αγοράς του Ηνωμένου Δεν θέλω να επικεντρωθώ πολύ στους δασμούς. Αυτό είναι θέμα της Τελωνιακής Ένωσης. Φυσικά και είναι σημαντικό στοιχείο η δασμή, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Εξαρτάται από τους κλάδους, από το επίπεδο των δασμών και εννοείται ότι χρειάζονται και υποδομές, έλεγχοι στα σύνορα προκειμένου να εφαρμοστεί ένα σύστημα με δασμούς. Αλλά αυτό είναι μέρος της εικόνας. Αυτό που έχει σημασία για την οικονομική ολοκλήρωση είναι πιστεύω η μη δασμολογική φραγμή σε σχέση με τη ρύθμιση της αγοράς. Οπότε για το Brexit εδώ έχουμε πολλές αβεβαιότητες. Στη μελέτη θέλησε επίσης να παρουσιάσω και τη σημασία που έχει και η σύνδεση με διάφορες πολιτικές, όχι μόνο του ανταγωνισμού, αλλά την περιβαλλοντική πολιτική, ακόμα και προστασία των καταναλωτών γιατί και εδώ τα δύο αυτά μοντέλα ολοκλήρωση της αγοράς, δηλαδή και απελευθέρωση του εμπορίου, εμφανίζονται εντελώ διαφορετικά. Ποιε είναι επίση κάποιε βασικέ αρχέ, η αμοιβαία αναγνώριση, για παράδειγμα, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα, εναρμόνιση. Αυτό είναι ο στόχο μου με τη μελέτη αυτή. Επίση, εγώ τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω τις διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα και τα δύο πρότυπα είναι προσοχή, mind the gap ή the gaps, τις διαφορές δηλαδή ανάμεσα ακριβώς αυτό που λέγαμε την ολοκλήρωση της αγοράς και την απελευθέρωση του εμπορίου. Αμοιβή αναγνώριση είναι ένα θέμα γιατί το Ρωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι θέλει σε βάθος και συνολικά συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ακόμα και να δεχτεί και τελωνική ένωση σε ένα βαθμό. Στα πλαίσια λοιπόν μια τέτοια συμφωνίας σε βάθος και εφόσον δεχτεί τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ιδέα είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα τότε αμοιβές αναγνώρισης. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν κόκκινες γραμμές που βάζει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν προσπαθείτε να δείτε τι υπάρχει στην αμοιβαία αναγνώριση και πώς αυτή λειτουργεί στην εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μιλάω εδώ πέρα για την συμμόρφωση που αποτελεί ένα μικρό μονομέρος της αμοιβαία αναγνώρισης, ενώ την αναγνώριση την αμοιβαία για κανονισμούς που αφορούν προϊόντα, ρυθμίσεις, μέσα από την εναρμόνιση της νομοθεσίας λειτουργεί η αμοιβαία αναγνώριση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι οδηγίες, πολύ περισσότερο από την ομολογία, οι οδηγίες οι ευρωπαϊκές που επιτρέπουν ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης και εξού και η αμοιβαία αναγνώριση. Άρα πλήρη συμμετοχή στο νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι η δυσκολία. Και στο ακαδημαϊκό επίπεδο ο κύριος Νικολαίδης, καθηγητής στην Οξφόρδη, έχει δημοσιεύσει στο blog του τις ευκαιρίες προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η αμοιβή αναγνώριση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλα πανεπιστήμια. ένα είναι πολιτικός αναλυτής, ο άλλος δικηγόρος, εγώ είμαι δικηγόρος, από αυτή την πλευρά μιλάω περισσότερο. Οπότε αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει πραγματικά να αποχωρήσει από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε η, πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να αποτελέσει μέρος της Βρετανικής Νομολογίας. Και δύο λόγια τώρα για τις υπηρεσίες πάλι θα σας δώσω μια προσωπική γνώμη. Αν τολμήσετε να συγκρίνετε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την απελευθέρωση του πορείου στον τομέα των υπηρεσιών, θα δείτε, νομίζω, πραγματικά, ότι η ιδέα να πετύχουμε απελευθέρωση διεθνούς εμπορίου μέσα από ένα ενοιολογικά ενωπημένο σύστημα που δημιουργήθηκε όταν δημιουργήθηκε ο ΠΟΕ με τις συμφωνίες γκάτσια, υπηρεσίες κλπ. για την εμπορία αγαθών, κατάργηση των εμποδίων, πρόσβαση στις αγορές, μη διάκριση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Απέτυχε στον ΠΟΕ και ακόμα και στις πιο προηγμένες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστα υπάρχουν όσον αφορά πραγματικά την απελευθέρωση του εμπορίου και των υπηρεσιών. Είναι κάτι υπηρεσίε και το εμπόριο δηλαδή που ναι μεν ε, έχουν ανοίξει πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απελευθέρωση μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες του ΠΟΕ περισσότερο τομεακά έχει συμβεί αυτό ή με νομοθεσία στο εσωτερικό επίπεδο. Συνεπώς, δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για τις υπηρεσίες. Έρχομαι τώρα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πιστεύω ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σαν μια μη οικονομική πολιτική, δεν μπορούμε να το δούμε ούτε μόνο από την οπτική γωνία της μετανάστευσης. Ε, συνεισφέρει στην ε, ολοκλήρωση βέβαια της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά είναι και πολύ πολιτικό το ζήτημα για το τι θα επιτρέψουμε και τι όχι αν θα επιτρέψουμε το άνοιγμα της αγοράς να αντισταθμιστεί από ευκαιρίες που θα δώσουμε στους ανθρώπους να εργαστούν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι σαν δικηγόρος θα αναφερθώ στα δύο επόμενα. Η απελευθέρωση του διεθνού εμπορίου λειτουργεί μέσω συμφωνιών που ενσωματώνονται στην διεθνή νομοθεσία. Δεν ε, αναγνωρίζεται η επιρροή του σώματος αυτού στο διεθνές εμπόριο. Ε, λέμε συχνά ότι το Brexit δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ το διεθνές εμπόριο. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ, αλλά πρόκειται για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί μέρος της εθνικής νομοθεσίας πια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η αόρατη πτυχή του εμπορίου και της ολοκλήρωσης που συχνά ξεχνάμε το γεγονός δηλαδή ότι η ολοκλήρωση είναι πραγματική εφόσον ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην Εθνική Νομοθεσία. Και άρα οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιοδήποτε εμπορεύεται μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια αποτελεσματικά για την εφαρμογή ακριβώς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υπάρχει η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπου υπάρχει πρόσβαση μέσω των εθνικών δικαστηρίων. Αν αυτό το συγκρίνεται με το τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, στον ΠΟΕ, ε, το όργανο ε, το οποίο ε, ξέρουμε, στο οποίο οι Αμερικανοί δεν ορίζουν νέα μέλη, το μποϊκοτάρουν, και τα συστήματα που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μελλοντικά συστήματα δεν λειτουργούν αρκετά καλά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια απόφαση που έχει αποφασιστεί από τέτοια όργανα ακόμα. Άρα παραμένουν μεγάλες διαφορές. Τώρα επειδή περνάει και ο χρόνος για τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες. Και εδώ πάλι η ολοκλήρωση της αγοράς έτσι όπως την ξέρουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απομακρύνεται περισσότερο από την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Και αυτό μέσα από τη δημιουργία οργανισμών που απαιτούν ρυθμιστικές εξουσίες. Δηλαδή, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράμε προς ένα σύστημα που θα ήταν ε, εκτελεστικό, ομοσπονδιακό και θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο μία χώρα μη μέλος να συμμετέχει σε ένα τέτοιο σύστημα και να δέχεται να αποτελεί μέρος της ένωμης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, κάτι που δεν υπάρχει στην ε, μελέτη είναι η εταιρική σχέση, η τελωνιακή εταιρική σχέση. Το Φεβρουάριο δεν φαινόταν η ιδέα αυτή να μπορεί να προχωρήσει από τις συζητήσεις που γινόντουσαν μεταξύ κυβερνήσεων εδώ, αλλά και πάλι φαίνεται να εγκαταλείπεται η ιδέα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάτι για αυτό που λέμε Customs ε, Partnership. Αυτό τι εννοεί, εννοεί κάτι σαν τελωνιακή ένωση. Αν όμως δούμε την εταιρική σχέση, θα ήταν ε, μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρούσε την εξουσία να έχει μια ανεξάρτητη εμπορική πολιτική και να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με οποιοδήποτε ανά τον κόσμο. Οπότε η ιδέα συλλογή δασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήδη τεχνικά δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά ακόμα και αν μπορούσε να λειτουργήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επέμενε για τους κανόνες προέλευσης που θα έπρεπε να τηρεί και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλιώ. το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να έχει εμπορικέ συμφωνίε που επιτρέπουν εισαγωγή ανταλλακτικών ε, αυτοκίνητα χωρί ε, δασμού και αυτό προφανώ μετά θα κυκλοφορούσε αυτά τα ανταλλακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον είχε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, τότε όμω θα είχε εμπορικό πλεονέκτημα. Οπότε εγώ δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια εταιρική σχέση τελωνιακή. τι θα μπορούσε να γίνει τώρα με τις εμπορικές συμφωνίες που έχει ήδη συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα το αφήσω για τη συζήτηση και συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα, ξεπέρασα το χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Αρκάουτ. Τώρα έχουμε 25 λεπτά περίπου για ερωτήσεις και απαντήσεις. Request floor. And who is the first? Ποιος ζήτησε πρώτος το λόγο. Ο κύριος Κάμπελ Μπένιμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον καθηγητή. Πολύ κατατοπιστική έκθεσή του και πολύ σωστή. Εγώ τι ήθελα να πω σχετικά. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Αυτά που προτιμούν οι Βρετανοί βασικά είναι ε, μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών τύπου ενισχυμένη, υπερενισχυμένη συμφωνία με Καναδά. Αυτά το πρότεινα στις 7 Μαρτίου, αλλά ε, εγώ προτείνω να καλύπτονται όλοι, όλοι οι τομείς με μηδενικές ε, ε, ρυθμίσεις, ε, δηλαδή μηδενικούς δασμούς, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, και να καλύπτει και τις υπηρεσίες όπως και οι υπόλοιπε συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών. Άρα έχουμε την υπερενισχυμένη ΣΕΤΑ που είναι καλή βάση ε, κατά την άποψή μου. Στις 13 Μαρτίου είπε ο κύριος Μπαρνιέ στη συζήτηση για το Brexit ότι τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη. Ο ΕΟΧ ή η Τελωνιακή Ένωση δεν νομίζω να είναι επιλογές και παραμένει η συζήτηση ε, και στη Βρετανική Βουλή 15 τροπολογίες ε, ε, τις οποίες η Βουλή των Κοινοτήτων μάλλον θα ανατρέψει. Θα παρακολουθείτε κι εσείς φαντάζομαι. Δεν νομίζω να ανατραπούν. Υπάρχει μεγάλη ε, ανησυχία του κόσμου και πίεση να σταματήσουν οι ολιγορίες και να προχωρήσουμε προς μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. γιατί επειδή γίνεται πολύ φασαρία και είναι γι' αυτό ασέβεια ε, προς το Βρετανικό λαό, θα πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε για τον ΠΟΕ, κύριε καθηγητά, και θέλω να σας ρωτήσω. Η μετάβαση μπορεί να γίνει αρκετά ομαλά στη σελίδα 24 της μελέτης σας. Με τα τελωνιακά τι γίνεται σε σχέση με τον ΠΟΕ. Ή θα χρειαστεί ειδική συμφωνία να συνεχιστούν οι σημερινές ε, τελωνιακές ρυθμίσεις μέχρι να υπάρξει κανονική οριστική συμφωνία ακόμα και υπό το πρίσμα του ΠΟΕ. Αυτά είναι τα κυριότερα που είχα να σας πω. Ευχαριστώ κυρία Μόσκα. Ε, Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια, διότι πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες ε, που ακούσαμε για τα θέματα αυτά. Επικροτώ λοιπόν ε, ε, τέτοιας μορφής υποστήριξη. Κάποια σκέψεις για τις προτάσεις που έγιναν. Από ό,τι μου φαίνεται ότι κατάλαβα από τη μελέτη, οποιαδήποτε λύση προτείνεται δεν επιλύει το πρόβλημα το οποίο συζητούμε συνεχώς, δηλαδή τη σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Στη μελέτη δεν διαπιστώνεται κάποια ε, δημιουργική λύση και καμία από τις πιθανές επιλογές ε, δεν καταφέρνει να δώσει τη σωστή άγουσα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση που είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο. Δεύτερο θέμα, στο οποίο θα ήθελα να ζητήσω περαιτέρω διευκρινήσεις, είναι το θέμα της δικαιοδοσίας. Διότι πράγματι υπάρχουν διάφορα επίπεδα αποδοχή των διαφόρων δικαιοδοσιών, αλλά από ό,τι μου φαίνεται κάθε επιλογή που προβλέπεται, είτε από τεχνικής είτε από πολιτικής σκοπιάς, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και τέλος, ε, κάτι τελευταίο, το οποίο ε, δεν ε, ε, εξήγησε πιο αναλυτικά λόγω έλλειψης χρόνου ο συντάκτης, πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον των εμπορικών συμφωνιών που αυτή τη στιγμή ισχύουν. το οποίο θεωρείται περιθωριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά μήπως στην πραγματικότητα οι εταίροι μας ε, θα μπορούσαν, ε, όπως κάνουν ήδη, να ε, θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ε, το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, ο Χέλμουτ Σόλ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο καθηγητή για την παρουσίασή του. Τρία σύντομα ερωτήματα την ομάδα παρακολούθησης του Brexit είχαμε ανταλλαγή απόψεων και για την Τελωνιακή Ένωση. Δεν υπάρχει εκεί καμία σαφήνεια έτσι, πολιτική, ούτε καν για το ποια κατεύθυνση θέλουμε να, να ακολουθήσουμε. Πολύ σκοτεινά. Ε, αυτά μεγάλη ομίχλη επικρατεί εκεί για ε, το τι θα γίνει μετά το Brexit και κρεμεί ακόμα και ε, το θέμα της ε, μεταβατικής περίοδου. Στη μελέτη σας αποφεύγετε κάπως να δώσετε και εσείς την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Τελικά τι σημαίνει αυτό. Αν δείτε την εσωτερική δομή κάποιων μονάδων παραγωγής Βρετανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπιστώσετε ότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής και αυτό ε, θα έχει επιπτώσεις στο κόστο του προϊόντος που μπορεί να είναι βρετανικό αλλά μπορεί να είναι και ευρωπαϊκό ανάλογα με τη δομή της επιχείρησης. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό και τι σημαίνει για το μέλλον των εμπορικών και παραγωγικών ε, προοπτικών βρετανικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι σημαίνει αυτό για τις θέσεις εργασίας και πώς θα επηρεαστούν. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στις υπηρεσίες και το σχετικό πρόβλημα. Από τη σκοπιά της απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Οι διαπραγματεύσεις ΤΙΖΑ γνωρίζουν επίσης δυσκολίες. Διότι οι υπηρεσίες θα επηρεαστούν όχι μόνο από την απελευθέρωσή τους, αλλά και από άλλα στοιχεία και από άλλες παραμέτρους. Οι εργαζόμενοι εκεί όσοι παρέχουν υπηρεσίες ε, θα επηρεαστούν από τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα οργανώσουμε στο μέλλον την ε, ανταλλαγή υπηρεσιών. Θα πρέπει να βρούμε και μια συμφωνία για το διαζύγιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Brexit και για τα δικαιώματα των πολιτών. Μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε πώς βλέπετε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον καθηγητή για τη μελέτη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεται το τελευταίο και θέλω να το διαβάσω γιατί είναι σημαντική η δήλωση. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό που το φαινόμενο Brexit χαρακτηρίστηκε από τέτοια σφοδρή απόρριψη του ρόλου του common law ε, στη Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση. Δηλαδή απορρίπτει ε, η Μεγάλη Βρετανία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θέλει να επιστρέψει στην εθνική δικαιοσύνη όπου κυριαρχούν κάποιες πολιτικές και κομματικές βλέψεις και όχι δημοκρατική διακυβέρνηση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και μου αρέσει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ακριβώς η δημοκρατική διαβούλευση για να βρούμε κοινέ λύσεις σε κοινά προβλήματα και να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική μας ισχύ ως μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για να επιτύχουμε τα καλύτερα για τους πολίτες μας και μια πιο δίκαιη εμπορική πολιτική ε, στον κόσμο. Είναι πολύ ισχυρό αυτό το συμπέρασμα και πολύ σημαντικό. Κάθε ανάλυση για τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit ε, δείχνει ότι θα υπάρξει ανετικός αντίκτυπος. Εγώ είμαι από τη βορειοανατολική Αγγλία, η οποία θα πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε μορφή Brexit. Γιατί έχουμε εμείς εμπορικό πλεόνασμα ε, σε αγαθά ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις υπηρεσίες έχει το Ηνωμένο Βασίλειο πλεόνασμα. Εξού και το σχόλιο που κάνατε εσείς κύριε καθηγητά ότι όλη η συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχείται μέχρι στιγμής από τα τελωνιακά. Και αυτό είναι λίγο διαστραμμένο διότι εντάξει έχουμε ε, κατασκευαστική βιομηχανία και είναι πάρα πολύ σημαντική και στην περιφερειακή μας οικονομία, τη δική μου περιφέρεια. Αλλά η βιομηχανική παραγωγή είναι μικρό ε, κλάσμα μόνο του συνόλου της Βρετανικής οικονομίας. Και αν δείτε τι διακυβεύεται εδώ για, στη συμφωνία Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών FTA δεν καλύπτει τις ανησυχίες ε, του κλάδου των υπηρεσιών. Και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα πρέπει να δούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τη δική σας πρόταση στη σελίδα 18. ένα είδος ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ενισχυμένου από μια συνολική τελωνιακή ένωση. Και το θέμα που θα τεθεί στο Λονδίνο και μας ενδιαφέρει και οι άποψή σα. είναι το εξή. Αν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχουν και οι άλλες χώρες του ΕΟΧ στη λήψη των αποφάσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τις βασικές της χώρες και σε ένα δεύτερο κύκλο ο ΕΟΧ ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και για την περιφέρεια μου και αντίστοιχες περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω για τη μελέτη και για την παρουσίασή της. Θα ήθελα ή δυνατόν να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε ό,τι όχι σχέση με τις ρυθμιστικές αποκλίσεις, διότι για πρώτη φορά ε, διότι μέχρι τώρα στις εμπορικές συμφωνίες προσπαθούμε να βρούμε λύση ε, για τους δασμολογικούς ε, φραγμούς και ρυθμίσεις, ενώ εδώ είμαστε στην αντίθετη περίπτωση. Ξεκινάμε από μια ολοκλήρωση και θα περάσουμε σε αποκλήσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο και πώς θα την ελέγξουμε αυτή την απόκληση και πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή η απόκληση η οποία θα υπάρξει με πάσα βεβαιότητα θα επηρεάσει το δυνατόν λιγότερο ε, αρνητικά το εμπόριο. Και δεύτερον, όσον αφορά ε, το επόμενο ερώτημά μου, για τους τελωνιακούς ελέγχους. Προφανώς ε, τη στιγμή κατά την οποία δυστυχώς ε, θα φύγει η Ευρωπαϊκή, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχουν τελωνιακοί έλεγχοι. Πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει ομογενοποίηση και οι καλύτεροι δυνατές συνθήκες ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον φραγμοί, κυρίως για το εμπόριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Ντάρτμουθ. Και μετά ο κύριος Ντέιβιτ ε, Κάμπελ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Θα μπορούσα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κάμπελ και να μιλήσω μετά. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, απλώς ε, μια ενημέρωση. Η Judith Curtin Darling επέστησε την προσοχή ε, μας στην τελευταία παράγραφο και φοβάμαι ότι η γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη έκθεση. Εσείς τη γράψατε αυτή την παράγραφο μόνο σας ή σας επηρέασε κάποιος άλλος εκεί στην τελευταία παράγραφη. Αν μπορείτε να με το διευκρινίσετε, θα σας είμαι ευγνώμων. Και τώρα ο κύριος Ντάρκμουθ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια βασικά στοιχεία θα ήθελα να σας διαβάσω που φαίνεται να μην περνούν καθόλου στην όλη συζήτηση και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη συζήτηση, αναφέρομαι σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και στο ίδιο το δημοψήφισμα. Κάτι πολύ απλό. Αν θέλεις να εξάγεις αγαθά σε μια άλλη χώρα, πρέπει να υπακούσει τους κανόνες αυτής της χώρας. Αν θέλεις να εξάγεις αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως κάνει η Γερμανία και μάλιστα σε τεράστιους όγκους και αξία, οι γερμανικές αυτοκίνητοβιομηχανίες πρέπει να τηρούν την Αμερικανική νομοθεσία. Γι' αυτό ε, βλέπετε ότι πολλές φορές ε, υπάρχει ε, κάποια εξήγηση που λέει ότι αυτό δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση στις ΗΠΑ. Ε, υπάρχουν δηλαδή κανόνες. Το θέμα είναι κατά πόσον οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύουν για όλες αυτές τις εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, από όλους αυτούς τους τομείς και κλάδους, ε, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες κλπ. που δεν εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε γενικές γραμμές το 12% είναι ε, εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αυτό το ποσοστό μειώνεται που σημαίνει ότι το 80% δεν εξάγεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα με την ενιαία αγορά, το πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Τζούντι ε, Κέρτον Darling, είναι ότι αν είσαι στην ενιαία αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το 88% και τις 100% που θα γίνει 90% σε μερικούς μήνες της Βρετανικής οικονομίας, που δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα υποχρεούται να επιβαρύνεται και είναι επιβάρηση με όλους τους ευρωπαϊκούς νόμους, κανόνες ε, και οδηγίες. Και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο εσείς μπορεί να πείτε ότι αξίζει τον κόπο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο, τον κόπο αλλά τουλάχιστον πρέπει να συζητηθεί, διότι ε, το παραβλέπουμε, το αγνοούμε συνεχώς. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τι κάνει μεταξύ άλλων. Είναι ότι επιβάλλει τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Αν είσαι στην ενιαία αγορά, τότε είσαι υπό την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορεί να είναι και καλό. Δεν ήξερα ότι ήταν ε, και τόσο σημαντικό, γιατί λέει εδώ και μια τελευταία παρατήρηση, πολύ σύντομα. Ε, ας με ε, συγχωρήσει ο Πρόεδρος. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διακεκριμένου συναδέλφου και πολύ εξέχοντα πρόεδρο και συζητάμε τα προβλήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται εμπορική συμφωνία για να μπορεί κάποιο να κάνει εμπόριο ε, και μάλιστα επικερδέ. Και μάλιστα, οι τρει μεγαλύτεροι εξαγωγοί προς τη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι, Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και η Ρωσία, δεν έχουν εμπορικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε οι 5 στους 10 ε, μεγαλύτερους, ούτε 11 στους 20 ε, μεγαλύτερους Δεν χρειάζεσαι λοιπόν σε εμπορία και νομίζω ότι η έκθεση βλέπει τα πράγματα από την άλλη πλευρά του τηλεσκοπίου. Θα έπρεπε να το βλέπετε ανάποδα, να κυρίσετε το τηλεσκόπιο από την άλλη. Πώς θα ήταν αν δεν υπήρχε εμπορική συμφωνία και ε, γινόταν εμπόρια βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά. Ο καθηγητής μάλλον τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με κάτι το οποίο ήταν προς το τέλος των ερωτήσεων. Έγραψα όλη αυτή την έκθεση μόνος μου. Και την τελευταία παράγραφο στα συμπεράσματα. Και σκέφτηκα και τη δομή των παραγράφων και υποστηρίζω την κάθε λέξη. Νομίζω και ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είπα ότι μια μετάβαση προς τον ΠΟΕ θα ήταν ε, άμεση ή κάτι αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι τώρα που είναι αυτό στην έκθεσή μου. Αλλά το θέμα είναι τι συνέπειες θα είχε αυτό για τα τελωνία. Η μετάβαση σε μια σχέση ΠΟΕ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου σημαίνει απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει πλήρης εξωτερικούς δασμούς ε, στις, ε, στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλιώς δεν τηρεί ε, την βασική αρχή του ΠΟΕ. Επομένως, απουσία Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ή Τελωνιακής Ένωσης θα πρέπει να ισχύουν οι πλήρεις δασμοί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στις εισαγωγές από την Κίνα ή τις Ηνωμένε Πολιτείε. Για να αναφερθώ σε δύο χώρες τις οποίες δεν έχουν και εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά το επίπεδο των δασμών θα ε, εξαρτηθεί από τους αντίστοιχους δασμούς σε κάθε κλάδο, αλλά θα αφορά οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης και Βασιλείου. Και νομίζω ότι αυτό προφανώς απαιτεί και ελέγχου στα σύνορα, όχι νόμου μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας, αλλά ε, και της υπόλοιπης επικράτειας. Τώρα, υπήρχε μια ερώτηση για τη Βόρεια Ιρλανδία και λέτε ότι στη μελέτη μου δεν έχουμε μια δημιουργική λύση. Το δέχομαι απολύτω. Φοβάμαι ότι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες με τις κόκκινες γραμμές ε, που έχει θέσει η αγγλική κυβέρνηση και αν θέλετε τις κόκκινες γραμμές ή τις διαχωριστικές γραμμές ε, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλετε ε, δεν, θα είναι και, δεν είναι και απόλυτα σαφές πώς θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι θέμα μόνο τελωνιακής ένωσης, είναι και κάτι το οποίο ε, προκύπτει και από το γεγονό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία είναι και οι στην, ε, στην ε, εσωτερική αγορά και επομένω δεν χρειάζονται σύνορα. Και γνωρίζουμε και από την ιστορία μα πόσα χρόνια χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει δυνατότητα να γίνεται εμπόριο μεταξύ κρατών μελών χωρί φυσικά σύνορα και ελέγχου στα σύνορα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρειάστηκε 10 χρόνια και 300 νομοθετήματα. Δεν ναι. μπορώ λοιπόν να διανοηθώ ότι θα, δεν θα υπάρχει σύνορο χωρίς ε, να υπάρχει, όπως λέει και στην έκθεσή μου, να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ της Τελωνιακής Ένωσης αλλά και των κανονισμών της εσωτερικής αγοράς μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχει ειδικό καθεστώ για τη Βόρεια Ιρλανδία ή να επεκτείνουμε αυτό το ειδικό καθεστώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μείνει με κάποιο τρόπο το Ηνωμένο Βασίλειο στην εσωτερική αγορά και στην Τελωνιακή Ένωση. Οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί κάποιου ελέγχου. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα των φυσικών συνόρων. Υπάρχουν τρόποι για να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε την ανάγκη για φυσικά σύνορα αλλά νομίζω κατά πάσα πιθανότητα στο Ιρλανδικό πλαίσιο και δεν είμαι και εμπειρογνώμων επί του θέματος ο βαθμός στον οποίο θα υπάρχει ολοκλήρωση ε, της οικονομίας μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας πηγαίνει πέραν των φυσικών συνόρων και των ελέγχων. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ένα αποτέλεσμα του Brexit που δεν θα ζημιώσει αυτή την κατάσταση, εκτός και αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση και την εσωτερική αγορά. Υπήρξε και μια ερώτηση για τα προβλήματα όσον αφορά τη δικαιοδοσία. Υποθέτω ότι αυτό αναφέρεται στην επίλυση διαφορών. Πολλά θα εξαρτηθούν εκεί από τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η μελλοντική σχέση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα αρχίσει κάποιος να εξετάζει τη συνεργασία και πέραν της συνεργασίας ε, κάποιες κοινέ ρυθμιστικές προσεγγίσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου χρειάζεται κάτι περισσότερο από την παραδοσιακή διαδικασία επίλυσης διαφορών που έχουμε σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερο από ένα πάνελ στο οποίο έχουν πρόσβαση οι δύο πλευρές. Ε, χρειάζεται ένα σύστημα στο οποίο θα εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ομοιόμορφα η νομοθεσία σε γενικές γραμμές. Και το έχουμε αυτό ε, στον ΕΟΧ μέσω του κώδικα ΕΖΕΣ ε, και θέλουμε και κάτι αντίστοιχο ε, στο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Για τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, δεν θεώρησα να το θεωρήσω περιθωριακό πρόβλημα αυτό. Αν ρωτάτε την άποψή μου γι' αυτό, και αυτό σχετίζεται και με άλλα σχόλια τα οποία έγιναν από τα μέλη εδώ, η φιλοδοξία του Ηνωμένου Βασιλείου να αναπτύξει δικιά του εξωτερική εμπορική πολιτική, στην πράξη θα πρέπει να ξεκινήσει ε, με το να προσπαθήσει να προλάβει αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη. Να προσπαθήσει δηλαδή να εξασφαλίσει ότι τα πλεονεκτήματα των ε, εμπορικών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που έχουν αυτή τη στιγμή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες δεν θα περιοριστούν. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια αγορά με αυτή που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ε, έδινα συμβουλές προς μια τρίτη χώρα που δεν δίνω, ε, το διευκρινίζω αυτό, θα τους ε, συμβούλευα να προσπαθήσουν να αποκομίσουν κάτι περισσότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι κατάφεραν να πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαφέ ότι αυτέ οι εμπορικέ συμφωνίε δεν μπορούν να συνεχιστούν. Οι τρίτε χώρε έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε ότι δεν μα δεσμεύει πλέον αυτή η συμφωνία. Σχόλιο εκτό μικροφώνου του κ. Ντάρτμουθ. Τι αποδεικτικά στοιχεία θέλετε. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις από τρίτες χώρες ήδη, οι οποίες θέλουν να εξετάσουν κάποιες πτυχές των ισχυρών συμφωνιών. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί και πολύ δύσκολα μπορούμε να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από αυτού. Δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα είναι περιφερειακό και ειλικρινά η ιδέα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκομίσει πάρα πολλά εάν αποκτήσει δικιά του εμπορική πολιτική ε, με βρίσκει ιδιαίτερα επιφυλακτικό. Πρέπει να μπορείς να προσφέρεις κάτι στο διεθνές εμπόριο ε, και το μέγεθος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τελωνιακοί δασμοί και πιθανές συνέπειε για τις επιχειρήσεις. Πραγματικά με ανησυχεί πολύ αυτό. Και με ανησυχεί υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο οικονομικό μοντέλο και οι οικονομολόγοι προσπάθησαν όσο μπορούν να διαμορφώσουν κάποια μοντέλα για τις πιθανές συνέπειες ε, ε, για τα διάφορα σενάρια του Brexit, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε νομίζω να αντιληφθεί το βαθμό στον οποίο μια ουσιαστική αλλαγή στους κανόνες του εμπορίου που θα σημαίνει αποχώρηση από την ε, Τελωνιακή Ένωση, διότι έγιναν επενδύσει ε, με το σκεπτικό ότι μπορεί ε, να εμπορευτεί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανταλλακτικά σου μπορεί να τα στέλνει οπουδήποτε, συνεχώ, χωρί ελέγχου ε, και να μπορεί να παραδίδει και έγκυρα τα προϊόντα. Το τι θα σημαίνει να αποχωρεί κάποιο από αυτό το σύστημα για τι επενδυτικέ αποφάσει των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να το αντιληφθούμε και ο ΠΟΕ έχει ως βασικούς τους στόχους μεταξύ άλλων στην επίλυση διαφορών και υπάρχει στη συμφωνία ε, την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα του εμπορικού συστήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τους οικονομολόγους ε, σήμερα και αυτή η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα απειλείται από μια τέτοια αλλαγή που δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα διαμορφωθεί. Πραγματικά λοιπόν με ανησυχεί. Για τις υπηρεσίες. Νομίζω πράγματι ότι η ιδέα της δεκαετίας του 90 ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το διεθνές εμπόριο και τις ε, υπηρεσίες μέσω ενός συγκεκριμένου μοντέλου απελευθέρωσης του εμπορίου δεν ισχύει πια, διότι το εμπόριο και οι υπηρεσίες δεν ε, ε, προστατεύονται καθαρά από προστατευτικά μέτρα όπως τελωνία και δασμούς, ε, δεν έχουμε πλέον φυσικά σύνορα, έχουμε πραγματικούς περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά. Και ο λόγος για τον οποίο μπορεί να γίνουν πολύ πιο δύσκολα αυτά είναι γιατί κάθε χώρα ρυθμίζει τις υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο. Και πρέπει αυτά να τα δούμε ε, σε κλαδικό επίπεδο, διότι οι μεταφορές, για παράδειγμα, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίε, υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, δεν είναι συγκρίσιμες. Ε, και δεν ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο και για ε, πολύ ε, καλούς λόγους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να δούμε ποιες είναι οι κοινέ αξίες και να εξασφαλίσουμε ότι η εσωτερική νομοθεσία θα αντανακλά αυτές τις κοινέ αξίες αν θέλουμε να έχουμε περαιτέρω απελευθέρωση. Και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι εντός της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε πλήρες ελεύθερο εμπόριο στις υπηρεσίες χωρίς ε, τη βαθύτερη ολοκλήρωση. Ε, και ε, φυσικά και τα δικαιώματα των πολιτών επίσης. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο το βλέπει αυτό σε διάφορες συζητήσεις, για παράδειγμα με την Ινδία για Συμφωνία Ελευθέρω Μπορείου. Η Ινδική κυβέρνηση θα επιμένει να έχει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες της και τους παρόχους υπηρεσιών και φυσικά αυτό έχει άμεση σχέση και με θέματα μετανάστευσης. για τον ΕΟΧ και τη Δηλωνιακή Ένωση και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν το έχω τονίσει αυτό πάρα πολύ στην έκθεση, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και ο ΕΟΧ είναι προβληματικός ε, στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε. Όταν δημιουργήθηκε, νομίζω ότι ήταν καλή απάντηση σε κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, αλλά υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δημοκρατίας ε, στον ΕΟΧ και πραγματικά διαρωτώ με κατά πόσον μπορούμε να δούμε πιο δημιουργικά μια ε, δευτέρου επίπεδου συμμετοχή ή μια σύνδεση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτούς τους κανονισμούς που εγκρίνονται τελικά από αυτές τις χώρες που συμμετέχουν στον ΕΟΧ. Υπάρχει πεδίο νομίζω για συνεργασία με αρκετές τρίτες χώρες για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Ρυθμιστικές αποκλήσεις, πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε και να έχουμε τις λιγότερο αρνητικές ε, συνέπειες. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να σταματήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ήθελα να πω όμως το εξή. Αν είναι λιγότερο ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν αριθμιστικέ αποκλήσει. γιατί φοβάμαι ότι δεν συμφωνώ με τον αξιότιμο συνάδελφο ότι ε, το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου είναι για την ε, ε, αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκρίνει όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλη αγορά και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ότι δεν χρειάζεται στην ουσία να πείσει οι τρίτες χώρες να συμμορφωθούν προς τους κανονισμούς της. Ε, οι επιχειρήσεις αυτό κάνουν διότι θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Το ξαναείδαμε αυτό το πράγμα, θα δούμε πόσες φορές θα το ξανασυζητήσουμε. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα, σημείο 13 και έχουμε 10 λεπτά μόνο γι' αυτό. Παρακαλώ. Για ποιο θέμα θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχω ένα διαδικαστικό. Βάσει ποιο άρθρο του κανονισμού. Τέλο πάντων, σύντομα. Θέλω να ζητήσω να έχουν οι συνάδελφοι την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, γιατί και η κυρία Ντάλ και ο κύριος Μάρτιν έχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούνε. Νομίζω ότι ε, έρχονται διάφορα νέα ζητήματα και δεν έχουμε την ευκαιρία πραγματικά να συνομιλήσουμε. Ε, ίσως να είναι ένα νέο προηγούμενο, να μπορούν οι μιλητές να φέρουν νέα στοιχεία στη συζήτηση. Πρόεδρος, πάντα υπάρχει περιορισμός χρόνου. Όλοι βέβαια προσπαθούν να μιλήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Πάντα είναι πρόβλημα αυτό. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε και άλλη συζήτηση για το Brexit ξανά και ξανά. Ωραία, 10 λεπτά λοιπόν τώρα έτσι. Δεν μου χρειάζονται 10, 2 λεπτά μου χρειάζονται μόνο. Η συμφωνία που συζητάμε σήμερα διαπραγματεύτηκε μετά την ε, προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την προσχώρηση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει την ελληνική της ε, ε, Ένωση και βάσει των κανόνων του ΠΟΕ η Κροατία πρέπει να κάνει διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ για να υπάρξουν προσαρμογές οι οποίες γίνονται με το εξωτερικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προσαρμοστεί η νέα χώρα στους κανόνες. Το ίδιο έγινε και ανάμεσα στην Κροατία και τη Νέα Ζηλανδία για την εισαγωγή διάφορων κρεάτων όπου οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υψηλότεροι από ό,τι ήταν της Κροατίας πριν την προσχώρησή της. Η αύξηση πρέπει να είναι αναλογική και έχουν επιτευχθεί συμφωνίες τώρα, παλιότερα με την Βραζιλία για παράδειγμα και έδωσε την έγκρισή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμφωνία αυτή με την Βραζιλία στις 18 Μαΐου που μας πέρασε. Τώρα, ξεκίνησε το Μάιο του 2017 η ιστορία αυτή και μονογράφηκε το Μάρτιο ε, που μας πέρασε. Υπάρχει αύξηση για τα βοηδή και για το προβατοειδή και τα εγωειδή, νοπά, διατηρημένα με πλήψή ψήξη κατάψυξη και αρχίζει να ισχύει η αύξηση αυτή, αλλά θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη και γι' αυτό ζητάω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα εξαιτία της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος. Ωραία. Οι σκιώδες εισηγητές δεν είναι εδώ. Ναι, θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της Καρολίνας. Ε, να σας πω ότι στηρίζουμε και εμείς αυτή την έκθεση. Ωραία. David Κάμπερμαν. Όχι, εντάξει, στηρίζουμε αυτή τη συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Άλντε. Δεν θέλει. Και εσεί συμφωνείτε. Ωραία. Άλλος, ο κύριος Μπούκνερ. Νομίζω ότι είναι σαφή η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Χέλμουτ. Δεν είναι εδώ ο συγκητής μα αλλά και εμεί συμφωνούμε. Η FDD. Δεν υπάρχουν σχόλια. Ωραία. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ζηρόμ από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να σημειώσω ότι πρόκειται για την τελευταία συμφωνία που θα έχουμε όσον αφορά την προσχώρηση της Κροατίας. Πλέον έχετε συνηθίσει τη διαδικασία αυτή και σας ευχαριστώ πολύ που συμφωνείτε, που δίνετε τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συμφωνία αυτή. Πρόεδρος, Ντάνιελ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό που καταλήγουμε σε αυτά τα θέματα τόσο γρήγορα. Η Κροατία είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, οπότε πρέπει να κλείνουν αυτοί οι φάκελοι πια. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, λέει ο Πρόεδρος, και εγώ χαίρομαι που όπως είπατε είναι μία από τι τελευταίε τέτοιε προσαρμογές που έχουμε μπροστά μας. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 23η Μαΐου στις 6 και θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας 20 Ιουνίου. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το σημείο και συνεχίζουμε αν και πήγαμε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Η ψηφοφορία θα αρχίσει ακριβώς στις 10. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε. Ώρα ψηφοφορίας. Check our voting card. Παρακαλώ να ελέγξουμε τις κάρτες μας. Hello, Please use your voting card. Σας παρακαλώ βάλτε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας στο μηχάνημα για να τσεκάρουμε τα μηχανήματα. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. λοιπόν της ηλεκτρονική ψηφοφορίας. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. εντάξει τώρα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε, έχει ζητηθεί το σημείο 15 να αναβληθεί η περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες το ζητούν, όχι επί της ουσίας, του περιεχομένου του συμβιβασμού, αλλά μπορώ να σας πω και ως πρόεδρος της Επιτροπής ότι το ζητώ και εγώ, γιατί έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή Εξωτερικών να βρούμε μια κοινή προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Και αυτό έχει ζητηθεί αναβολή της ψηφοφορίας. Είναι το περίφημο άρθρο 53 συν. Εμείς είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας αλλά σε στενή επαφή και συνεργασία με τους αδέρφους της Επιτροπής Εξωτερικών, ΑΦΕΤ. Επίσης, ο κύριος Μακαλιστέρη είναι στην Σόφια και έχει χάσει και το κινητό του και τα λοιπά και δεν μπορούμε να τον βρούμε. <laughs> Χτες το έστειλα ένα mail και μου είπε ότι δεν συμφωνεί με το συμβιβασμό. Οπότε η πρόταση είναι να αυληθεί η ε, ψηφοφορία για τις 28 Μαΐου. Με ένα σαφές μήνυμα ότι εμείς ως Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε με το συμβιβασμό και με τη δήλωση για να τα διαβιβάσουν αυτά στους συναδέλφους Επιτροπής ε, ΑΦΕΤ. Πριν ψηφίσουμε αυτό το θέμα της αναβολής ψηφοφορίας για το σημείο 15, θα ήθελα να δώσω λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Βαλένσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα προτιμούσα να ψηφίσουμε σήμερα, διότι η αναβολή δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Έχουμε κατάλογο ψηφοφορία, έχουμε τη συμφωνία μεταξύ μα εδώ, ε, οι συνάδελφοι τη Επιτροπή μα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες τώρα να αναβληθεί για τις 28 Μαΐου τι θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Έχουμε μια άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβαστική πρόταση 1, τη λεγόμενη κοινή δήλωση που έρχεται να αντικαταστήσει πολλές ε, από τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει δικά μας μέλη. Και στο πνεύμα της καλής συνεργασίας έχουμε συμπεριλάβει και πολλές ανησυχίες και μελήματα της Επιτροπής Εξωτερικών. Δύο πράγματα είναι αυτά που δεν έχουν συμπεριληφθεί γιατί δεν συμφωνήσαμε ε, οι συνομοθέτες. Η πρόταση λοιπόν είναι πολύ καλή. Είναι καλή η συνεργασία που είχαμε με τους και ηγητές μου και είμαι πάρα πολύ ε, ευγνώμων για την κατανόησή τους και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Ωραία, σαφέ μήνυμα από τον εισηγητή. Αλλά θυμηθείτε ότι έχουμε και αυτή τη συμφωνία με την Επιτροπή Εξωτερικών. Παρ' όλα αυτά, εσεί θα αποφασίσετε αν θέλετε αναβολή τη ψηφοφορία ή να γίνει σήμερα. Έτσι λέει ο κανονισμό. Λοιπόν, ψηφίζουμε γι' αυτό ακριβώ το θέμα αν θέλετε να αναβληθεί όχι η να γινει σημερα ετσι λεει ο κανονισμο λοιπον ψηφιζουμε γι αυτο ακριβω το θεμα αν θελετε να αναβληθει η οχι η ψηφοφορια για το θέμα 15. Αν ψηφίσετε ναι, σημαίνει ναι στην αναβολή. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Άρα θα ψηφίσουμε σήμερα. So, point 14. Σημείο 14. Vote on uh, the TDI modernization. 14. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μία ενιαία άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping και επιδετούσαν εκ μέρου χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρας ψηφοφορίας. Με σαφής πλειοψηφία υπέρ εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο σημείο 15. Περαιτέρω μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 25 υπε. κατά αποχές απορρίπτεται ο έλεγχος φωνάζει ο κύριος Dartmouth αρχίζει βεβαίως η ηλεκτρονική επαλήθευση πέρασε Σαφέστατα έχει απορριφθεί, κύριε συντάκτα, της τροπολογίας. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής άφετη τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 6 καταπίπτει, 7 της Επιτροπής Εξωτερικών. Τα δύο εκρεμή ζητήματα ε, και τα πιο επίμαχα θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Το CND είναι αυτό η παράγραφη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 ε, της ΑΦΕΤ. Α, όχι, 8 καταπίπτει τώρα. Μετά η τρία της Επιτροπής Εξωτερικών έχει αποσυρθεί. Όχι, έχει αποσυρθεί 23. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. closed. Και τελειώνει. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Βαλένσα. Σημείο 16. Δημόσιες συμβάσεις και αντίστοιχη στρατηγική. Είναι του κυρίου Κασπάρη η έκθεση. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Α, όχι. Η επιτροπολογία 5, το δεύτερο τμήμα, διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τοπολογία 8 προς τα εκεί κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται και συγχαρητήρια Ντάνιελ Κασπάρη. Λήξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και προχωρούμε. Στο σημείο 18. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ, ο οποίος θα αναλάβει να προεδρεύσει ε, για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Καλή συνέχεια και καλά να περάσετε μέχρι την επόμενη φορά. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν, να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση αυτή, να αποχωρήσουν ησύχω. Πάμε στο σημείο 17, λέει ο Πρόεδρος. Αντιπροσωπεία ad hoc στην Κίνα. 7 με 9 Μαΐου 2018. Πήγαμε στη Σανγκάη και εκεί συναντηθήκαμε με την ε, πρόεδρο του Κογκρέσου εκεί και μείναμε και στο Πεκίνο δύο μέρες όπου συναντηθήκαμε με διάφορους υψηλά ιστάμενους ε, υπεύθυνου για αποφάσεις, τον Υπουργό Εμπορίου, τον ε, επικεφαλής του Κινέζικου Κογκρέσου και τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής εκεί. Συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους δύο σημαντικών ε, σωμάτων. Το ένα είναι η Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης, που είναι η υπεύθυνη για την κατάρτιση της οικονομικής πολιτικής και το άλλο σώμα ήταν το υπεύθυνο για τη ρύθμιση των αγορών κάτι για το οποίο ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Ε, δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή μετά από την προσπάθεια μεταρρυθμίσεων κλπ. Η αρχή αυτή είναι ένα νέο όργανο όπου συμμετέχουν διάφορες ρυθμιστικές αρχές κατά το παρελθόν και τώρα έχουν συγχωνευτεί όλες μαζί. Η αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε και με εκπροσώπους ε, ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. Μα πού είναι το σφυρί μου. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, ησυχία. Ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με το εμπορικό επιμελητήριο στην Κίνα, τόσο στο Πεκίνο όσο και στη Σαγκάη. Όπως ξέρετε, το επιμελητήριο αυτό είναι εταίρος της δικιάς μας Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και συστήσαμε και την επόμενη συνάντησή μας όταν θα έρθουν το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες. Θεωρώ ότι ήταν πολύ επικαιρή η συνάντηση αυτή γιατί δεδομένων των μονομερών αποφάσεων πολλές φορές πλήττεται και το εμπόριο. Συζητήσαμε λοιπόν και επιμείναμε στη στήριξή μας του πολυμερούς, στο πολυμερές σύστημα και με τους Κινέζους είπαμε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις που να είναι συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ πιέζουμε να ολοκληρωθεί και συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την συνολική ε, συμφωνία για τις επενδύσεις. Ακούσαμε πολλές πολιτικές δεσμεύσεις. Ανακοινώθηκε το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας οικονομικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων και γενικότερα όσον αφορά την ε, εφαρμογή νέων μέτρων. Ήταν μια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε και τις διαφορές που υπάρχουν από τους εκπροσώπους των κομμάτων αφενός που ήταν πιο φιλόδοξες και τις λιγότερο φιλόδοξες ε, δηλώσεις για παράδειγμα του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας. Τώρα οι συμμετέχοντες από τους σοσιαλιστές ο Ντέιβιτ Μάρτιν, αν έχει να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας ευχαριστώ τη Γραμματεία για την οργάνωση της αποστολής αυτής. Ήταν πολύ καλή. Συναντηθήκαμε πράγματι με τους περισσότερους ανθρώπους ε, τους οποίους επιθυμούσαμε και να συναντήσουμε σύντομα τώρα μετά από τις δικές σας, τα δικά σας σχόλια για τις γεωγραφικές ενδείξεις υπάρχει μια ελπίδα. Οι Κινέζοι να προχωρήσουν και να υπάρξει συμφωνία. Έχουμε τη διάσκεψη κορυφής τον Ιούλιο, δεν νομίζω πριν από αυτό να γίνει. Από την άλλη όμως ε, πιέζεται η Κίνα και για τη συμφωνία όσον αφορά τις επενδύσεις. Εκεί δεν είδα ισχυρή βούληση. Δεν ξέρω και αν κατάλαβαν τις επικρίσεις μας για την έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά τους εμπορικούς κανόνες. Τι γίνεται δηλαδή με τους Ευρωπαίους επενδυτές στην Κίνα σε σχέση με αυτό που γίνεται για τους Κινέζους επενδυτές στην Ευρώπη δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ε, ήταν πολύ συμπαθείς, μιλήσανε για αλλαγέ, αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι θα συνεχίσουν. Οπότε τη δικιά τους ε, την πλευρά θα συνεχίσουν να προστατεύουν βέβαια τα κινέζικα συμφέροντα. Και το πιο ενδιαφέρον ήταν από τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες που είπαν το θέμα των σχέσεών μας με την Κίνα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι κινέζικο. Οπότε εμεί θα έπρεπε να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι. Οι Κινέζοι σέβονται ότι κάνουμε εφόσον προχωρήσουμε με τις προτάσεις μας για τον αμυντικό μηχανισμό, οι Κινέζοι μας σέβονται γι' αυτό. Και αν θέλουμε να αλλάξει η ισορροπία, Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα γίνει εφόσον η Ευρώπη θα είναι αποφασιστική και επίμονη σε αυτά που θέλει να ζητήσει από τους Κινέζους. Ευχαριστούμε. Ο Σαλβατόρε Τσίκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω καταρχάς και να δώσω συγχαρητήρια για την πάρα πολύ αποτελεσματική οργάνωση αλλά επίσης ε, και να συγχαρώ μια αντιπροσωπεία η οποία με πολύ ισχυρό τρόπο και αποφασιστικό τρόπο κατάφερε να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ταυτότητα ενός κοινοβουλίου που σε εκείνο το πλαίσιο ε, ήρθε να ε, ε συζητήσει με την κινέζικη πλευρά. Ε, νομίζω ότι καταφέραμε να εμβαθύνουμε αρκετά όλα τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και επίσης νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε κάποια επιρροή για τον Ιούλιο που πιστεύω ότι θα μπορούσε να καθορίσει την πιθανή και εγώ ελπίζω συγκεκριμένη συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επίσης είδαμε και με ποιο τρόπο η Κίνα χρειάζεται στην ε, ιδέα της ε, μια ιδέα 30 ετών με μεταρρυθμίσεις ε, που οδήγησαν το Κογκρέσο της και την Εθνοσυνέλευση να έχει ένα προγραμματισμό και να ασχολείται και με την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένους όρους. Επομένως, πίστηκα ότι από αυτή την συζήτηση, την συνάντηση υπάρχει ανάγκη και από δικής μας πλευράς να δούμε ε, τι ακριβώς κάνουν. Ε, ε, θέλουν να φτάσουν σε μία διάσταση η οποία πηγαίνει πέραν των σχέσεων που έχουμε με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και επίσης μία ακόμα πτυχή. Εμείς πήγαμε εκεί σε μία στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία παγκόσμια διεθνής κατάσταση που όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και το σύστημα μέσω των θέσεων του Προέδρου Τραμπ και το παγκόσμιο σύστημα το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ θέλει, αν θέλετε, να επανεκκινήσει ε, και με κάποιο τρόπο να ρυθμίσει βάσει του δικού του ε, προγράμματος και είναι προφανές ότι η δική μας αντιπροσωπεία βρέθηκε να κάνει ε, αξιολογήσεις αντιπαράθεση αυτού του τύπου διότι ενώ εμείς συζητούσαμε με την αντιπροσωπεία και τα διάφορα ε, σημαντικά επίπεδα της Κίνας οι κοινωνικές αντιπροσωπείες μιλούσαν και με την αμερικανική αντιπροσωπεία και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ απλώς σε αυτό το οποίο γνωρίζετε ότι συνέβη για μία από τις μεγαλύτερες ε, κινέζικες επιχειρήσεις, τη Z, για την ε, ε, επιβολή των δασμών, η οποία αποσύρθηκε από πλευρά Τραμπ και αποσύρθηκε ακριβώς τις ημέρες που εμείς ήμασταν στην Κίνα και συζητούσαμε τις συμφωνίες μας και την απέσυρε, διότι οι συζητήσεις αυτές μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων οδηγούν σε πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες, οι οποίες αναπόφευκτα αφορούν και μας. Και μάλιστα εγώ σήμερα το πρωί ε, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον μια ανταλλαγή απόψεων και είναι προφανές ότι ο Τραμπ δημιουργεί συμμάχους, κυρίως με την Κίνα, αλλά δημιουργεί και συμμάχους ε, και με την Κίνα για το παιχνίδι το οποίο παίστηκε και με τη Βόρεια Κορέα. Ε, επομένως εμείς σε αυτό το πλαίσιο κάναμε μια αξιολόγηση και μια απελήθευση που πηγαίνει πολύ πέραν τη απλή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Και φυσικά συγχαρητήρια και σε εσά κύριε Πρόεδρε που είστε ο μόνιμο εισηγητής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα, ο κύριο Βινκλέρ, ο οποίο κατάφερε ε, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα να προχωρήσει αυτό το διάλογο, τον οποίο σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ιδιαίτερο θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σχάκη. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά υπόθηκαν ήδη, αλλά να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή, η πρώτη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και ελπίζω όχι τελευταία. Μας υποδέχτηκαν σε υψηλότατο επίπεδο. Είχαμε ειλικρινείς συζητήσει, αν και μερικές φορές ε, χαθήκαμε πραγματικά στη μετάφραση, κυριολεκτικά. Χρειάζεται χρόνος. Το βασικό πάντως που περιμέναμε ήταν μια προσέγγιση βάσει κανόνων και αυτό το καταστήσαμε σαφές επικεντρωθήκαμε στο πρόβλημα της υπερικανότητας ε, εξαγωγών της Κίνας, ε, στην τήρηση των κανόνων και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία έχει μπροστά της η επιχειρηματική κοινότητα. Μας τα εξήγησαν διακρίσεις, ε, dumping, ακόμα και αν δεν είναι γραμμένα άσπρο-μαύρο, υπάρχουν. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε μια συνολική στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα που να μην ασχολείται μόνο με τα θέματα της δικιάς μας Επιτροπής αλλά με τις ψηφιακές εξελίξεις, την ε, ε, τεχνητή ευφυΐα, ε, διάφορα άλλα πρωτοβουλίες, ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε ολόκληρη μερίσια διάταξη για τέτοια ζητήματα που να συμπεριλάβουμε σε μια τέτοια στρατηγική. Μιλήσαμε σύντομα και για το ψηφιακό εμπόριο, που σίγουρα είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε για να καταπολεμιστεί ο προστατευτισμός και άλλοι περιορισμοί που μπαίνουν από την Κίνα στην Ευρώπη. Αυτά που ακούσαμε ήταν ε, λογικά για το εμπόριο βάση κανόνων, για παράδειγμα. Αυτά τα ακούσαμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι και η πρακτική που ακολουθεί η Κίνα ε, ευθυγραμμίζεται στα λόγια τους. Οπότε μπορεί να τίθεται και λίγο θέμα αξιοπιστίας ακόμα και αν ήταν πολύ καλό που πήγαμε και μιλήσαμε εκπροσώπους της κυβέρνησης αλλά και άλλους στο Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο για να καταλάβουμε κατά πόσα αυτά τα οποία υπόσχονται όντως γίνονται και στην πράξη. Εκεί λοιπόν βάζω ένα ερωτηματικό καταρχήν. Αυτά προς το παρόν και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε για πολύ στο θέμα αυτό της Κίνας για να είναι ξεκάθαρο το τι περιμένουμε από αυτούς. Ευχαριστούμε. άλλο κανεί Σχόλιο. Α, παρακαλώ, κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ για την ε, παρουσίαση αυτή όσον αφορά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Κίνα. Εγώ αναρωτιέμαι και δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να απαντήσετε τρεις ερωτήσεις για την αντιπροσωπεία αυτή. Υπήρχε διμερής αντιπροσωπεία Κίνα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τι βαθμό είχατε την ευκαιρία να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο για τις μελλοντικέ σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας στις συνομιλίες που αναφέρατε. Δεύτερον, είπατε είχατε επαφές υψηλού επίπεδου στο πρόγραμμα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κίνα σε τι βαθμό έπαιξε ρόλο στις συζητήσεις που είχατε. Αναφέρθηκε καθόλου αυτή η έκθεση σε σχέση με τις επιδοτήσεις, ε, τους εμπορικούς περιορισμούς κλπ. που επιβάλλουν οι Κινέζοι. Και τέλος, στην τελευταία συνέλευση του ΠΟΕ, οι Κινέζοι δεν ήταν παρόντες. Μετά την κοινοβουλευτική συνέλευση αυτή, λοιπόν, στο Buenos Aires, καταλάβαμε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί η συνεργασία με την κινέζικη πλευρά. Με μέλη δηλαδή του Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας. Ακούσαμε για τις δεμερείς σχέσεις Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε ότι συζητήσατε για αυτά. Εγώ θέλω να ξέρω η απροθυμία των Κινέζων να, να συμπεριλάβουν το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε συμφωνίες η συμμετοχή τους και με ποιο τρόπο σε εμπορικές σχέσεις είναι πράγματα που συζητήθηκα. Προσπαθήσατε να βρείτε δηλαδή μια νέα προσέγγιση στη συνεργασία μας με την ε, Κίνα και τους κοινοβουλευτικούς, γιατί και εμείς πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Θα προσπαθήσω λίγο να απαντήσω και να κάνω και ένα σχόλιο ε, από πλευράς μου, όχι ως πρόεδρος, αλλά ως εισηγητής για την Κίνα. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις σου, Χέλμουτ. Η πρώτη είναι μια ερώτηση που πραγματικά ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι αν απαντούσα απευθεία στην ερώτησή σου, θα πρέπει να πω ότι οι επισκέψει μα ήταν συμπληρωματικέ με την αντιπροσωπεία τη Κίνα. Δεν υπήρχε καμία αλληλοεπικάλυψη και δεν ε, συντονιστήκαμε ή δεν αναλύσαμε ε, τις εντολές μας, αλλά ήταν συμπληρωματικές επισκέψεις. Και τώρα, και εδώ έχετε η προσωπική μου άποψη, ε, πιστεύω και αυτό θα ήθελα να το προτείνω κιόλα ε, για μία από τις επόμενες συνεδριάσεις ε, των συντονιστών εδώ στην Επιτροπή και στην ηγεσία της Επιτροπής, και να το επισημάνουμε ίσως και στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, διότι δεν νομίζω ότι είναι επικοδομητικό να υπάρχουν δύο αντιπροσωπείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πηγαίνουν ταυτόχρονα στην ίδια χώρα. Δεν οδηγεί πουθενά και από ό,τι κατάλαβα, μία από τις επόμενες αντιπροσωπεία μας να αντιμετωπίσει μια ίδια κατάσταση. Θα πάμε στην ίδια χώρα με μία άλλη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω ότι είναι μεγάλο το Κοινοβούλιο και αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία των μελών και των επιτροπών να αποφασίζουν, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής ε, δεν θεωρώ ότι ωφελεί για τα συνολικά συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πηγαίνουμε στην ίδια χώρα, το ίδιο διάστημα, την ίδια εβδομάδα και να ε, στέλνουμε μηνύματα τα οποία επικεντρώνονται σε τελείως διαφορετικά θέματα και διαφορετικούς τομείς, διότι ο καθένας από εμά έχουμε τον τομέα μας. Αν μπορούμε λοιπόν να το σημειώσουμε και να συζητηθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσει των συντονιστών και να επισημοποιηθεί κάπως. Όχι, δεν άκουσα καμία αναφορά στις εκθέσεις αναχώρα, αλλά συζητήσαμε ε, τα θέματα που συζητήσατε, τις διαφορές ε, των εμπορικών μέσων και τις επιδοτήσεις. Η Κίνα από τη μια μεριά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα όσα συμβαίνουν για τις νομικές εξελίξεις και το έθιξαν αυτό και το έθιξαν και οι συνάδελφοι. Τι νομικές εξελίξεις ακούν ότι γίνονται, υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μηχανισμό επενδύσεων, για τα διάφορα ε, μέσα ε, προστασίας του εμπορίου κλπ. Αλλά από την άλλη υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις ε, για επιδοτήσεις και ενισχύσεις και υπερβολική παραγωγή. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν κυρίως στις πολιτικές συναντήσεις και δεν διαφάνηκαν τόσο σαφώς στο πιο ε, τεχνικό επίπεδο, αν θέλετε. Ε, είχαμε και κάποια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε κάποια στοιχεία μετά από τη συνεδρίαση στο Βερολίνο του Παγκοσμίου Φόρουμ για τις υπερβολικές παραγωγές ε, αλλά υπάρχει δυνατότητα να επαληθεύσουμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε αν αντανακλούν ή όχι την πραγματικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά το χάλιβα, ε, διότι είναι πολύ περίπλοκη η πραγματικότητα επιτόπου στην Κίνα και είναι πολύ μακρά ιστορία να καταλάβουμε πώς η υπερβολική παραγωγή σε τομείς που είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί ε, σταματά και κλείνει η παραγωγή και ε, ανοίγουν καινούργια σε άλλους τομείς. τώρα, για το θέμα του ΠΟΕ, Νομίζω ότι μπορώ να επαναλάβω την απάντηση που έδωσα και στην προηγούμενη ερώτηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δηλώσεις, αλλά οι δηλώσεις και τα στοιχεία δεν ε, συνάδουν μεταξύ τους. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ε, παρουσίας της Κίνας στον ΠΟΕ είναι κατά πόσον ασχολούμαστε με μια αναπτυγμένη χώρα ή με μια αναπτυσσόμενη χώρα και νομίζω ότι η νομοθεσία στον ΠΟΕ ε, είναι πολύ ανοιχτή ε, για αυτή την τόσο σαφή διάκριση, αλλά και αυτοί παίζουν πολύ άξιμα το παιχνίδι τους και φυσικά το επιχείρημα έρχεται λόγω του μεγέθους τους. Ε, διότι αν πείτε ότι το ένα τμήμα της παράκτιας Κίνας είναι αναπτυγμένο, αλλά στη Δύση και στο Βορρά έχουμε περίπου πληθυσμούς που είναι περίπου η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερη δηλαδή από οποιαδήποτε χώρα των Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, έχουν τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Έχουν και αυτοί κάποιο δίκιο, έχουμε και εμεί το δίκιο μας, αλλά ε, ο ΠΟΕ, επειδή ακριβώς ε, δεν είναι απόλυτα σαφή επ' αυτού, δίνει ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα σε αυτού και όχι σε εμά. Και ίσως, αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, θα μπορούσα να κάνω και μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να συζητηθεί και στο μέλλον για την Επιτροπή μας και τη σχέση μας με τους ε, Κινέζους εταίρους μας. Ναι, είναι τεράστια χώρα, αλλά αν μπορούσαμε να έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο να έχουμε τουλάχιστον επαφές μια φορά το χρόνο μία στις Βρυξέλλες, μία στην Κίνα. Ίσως θα ήταν ένας τρόπος να χτίσουμε και κάτι, γιατί αλλιώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, πηγαίνει στην Κίνα, μία ή άλλη επιτροπή πηγαίνει στην Κίνα κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και δεν συζητούν πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν εμάς. Επομένως, ε, ίσως θα μπορούσαμε να θίξουμε και αυτό το θέμα ε, σε κάποια επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Υπάρχει δυνατότητα να καλούμε και τους ε, Κινέζους εταίρους να έρχονται στις Βρυξέλλες Βρυξέλλες για διάλογο εξειδικευμένους, ε, το Υπουργείο Εμπορίου ε, ή κάποιους εμπειρογνώμονες και... Ε, να γίνεται ίσως και σε την ίδια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διάλογο με την Κίνα, να μπορεί να συμμετέχει η Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται νομικό σε αυτό, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε κατά πόσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ε, τέλος, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους αδέλφους που ευχαρίστησαν τη γραμματεία για τη δουλειά και την προετοιμασία. Ε, τα πάντα ε, πήγαν ομαλά και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Αν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο, να ολοκληρώσουμε με αυτό το σημείο. Επόμενο, σημείο 18, η δραστηριότητα των ε, ομάδων δραστηριοτήτων η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων, συγγνώμη, και εδώ έχουμε την ομάδα για την Ιαπωνία. Αυτή η ομάδα παρακολούθησης ε, προσπάθησε να ενισχύσει ε, τις εργασίες της για να προχωρήσει την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Ξέρετε ότι θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σύντομα για την συγκατάθεσή του. Συναντήθηκαν δύο φορές η συνάδελφος Σίλβα, ο συνάδελφος Σίλβα Περέιρα δεν είναι εδώ. Θα διαβάσω λοιπόν κάποιες σημειώσεις του. 25 και Απριλίου και 15 Μαΐου έγιναν ανταλλαγές απόψεων με ενδιαφερομένους Ευρωπαίους, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αυτοκινητοβιομηχανιών, ε, ε, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις μεταφορών και περιβάλλοντος και άλλους και οι Ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη συμφωνία. Κάποιοι άλλοι επεσήμαναν τα πιθανά ωφέλη μιας συμφωνίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, αλλά υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά ε, για παράδειγμα κάποιες εκκρεμείς κυρώσεις ε, δύο από των βασικών, εκ των βασικών συμβάσεων του Διεθνούς Διευθυντή ε, τα μη δασμολογικά μέτρα πρέπει να συζητηθούν επίσης στη συμφωνία και χρειάζεται περαιτέρω ευθυγράμμιση με διεθνή πρότυπα από πλευρά Ιαπωνία. Κρεμούν κάποια θέματα για την πλήρη απολευθέρηση των, του ευρωπαϊκού τομέα αυτοκινήτων και κάποια θέματα ευελιξίας και διαφάνειας που αφορούν τους κανόνες καταγωγής. εκφράστηκαν και κάποιες ανησυχίες ε, για τα παραδοτέα στο κεφάλαιο ε, του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης η Ένωση Τροφίμων και Ποτών ε, Ευρώπης ε, είπε ότι η Ιαπωνία είναι ε, κατά 90% αυτάρκης για τρόφιμα και επομένως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ενδιαφέρονται για εισαγωγές και θα ζητούν υψηλές απαιτήσει όπως αυτές που έχουν και οι ίδιοι. Οι συζητήσεις έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις πληροφορίες και να εξηγήσουν και κάποια αποτελέσματα. Στη συνέχεια έχουμε το Μεξικό. 25 Απριλίου η ομάδα παρακολούθησης για το Μεξικό συναντήθηκε με την Έλενα Κένινγκ, την διαπραγματευτή, για να συζητήσει ε, το θέμα του τμήματος του εμπορίου της εξυγχρονισμένης συμφωνίας και έχουμε τη μόνιμη συγγήτρια, την Μακολάδα Ροντρίγεθ Πινέρο και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να σας ενημερώσω. Εχθές μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Κιόνικ, προηγουμένως είχε ενημερώσει και την ομάδα παρακολούθησης, δεν είχε περισσότερες πληροφορίε. Ε, οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ ε, για την πληροφορία αυτή, για την ενημέρωση, έκαναν ερωτήσεις, απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Έχουμε και την ομάδα παρακολούθησης ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες που συζήτησαν με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου περιορισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για το χάλιβα και τον άνθρακα και το αλουμίνιο, συγγνώμη. δεν είναι εδώ ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Και τι να κάνουμε τώρα, να τον αναβάλουμε. Από πού είναι ο Βίγκλερ. Ε, υπήρξε κάποια ενημέρωση, αλλά όπως βλέπετε αλλάζει η κατάσταση από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αν δεν είναι εδώ ο αρμόδιος, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ για την Κίνα. Έχουμε, είχαμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου για το θέμα αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, διότι η ανταλλαγή αυτή απόψεων έγινε πριν την αντιπροσωπεία στην Κίνα, πριν την επίσκεψη εκεί της αποστολής και αφορούσε τη κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τη διμερή επενδυτική συμφωνία. Ουσιαστικά η ενημέρωση που μας έγινε εκεί αφορούσε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων και προετοιμασία του επόμενου γύρου. the Chinese uh, ε, οι Κινέζοι ε, εταίροι μας πολλές φορές έτσι παίζουν τις καθυστερήσεις και κολυσιεργούν γιατί δεν βιάζονται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Επίσης προβλέπεται ε, για το καλοκαίρι τον Ιούλιο, αν δεν απατώμε, σύνδρος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας αλλά προβλέπεται έτσι, δεν ξέρω. Είναι κάπως συγκρατημένη η αισιοδοξία και η φιλοδοξία για το τι θα γίνει. Γιατί η τελευταία σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ήταν ατελέσφορη. Μικρά, πενιχρά τα αποτελέσματα μόνο. Αυτά. Ουσιαστικά. Ήταν όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, ομάδα παρακολούθησης. Επόμενο θέμα, ε, Ηνωμένο Βασίλειο και Brexit και αντίστοιχη ομάδα παρακολούθησης. 15 Μαΐου συνεδρίασε αυτή και είχε ανταλλαγή απόψεων για την τελωνιακή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πάμπριξ είναι εδώ, ο μόνιμος εισηγητής μας και το δίνω το λόγο. Αυτή τη στιγμή αντικαθιστώ την Κοντελίβε Ρόβολ, και πραγματικά την τρίτη που μας πέρασε στην ομάδα παρακολούθησης για το Brexit ασχοληθήκαμε με τη μελλοντική πιθανή τελωνιακή συνεργασία μας. Πάρα πολύ σύντομα να πω για τους συναδέλφους ότι στην αρχή θέλαμε να προσκαλέσουμε ε, εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίων οι οποίοι αρνούνται να έρθουν γιατί λέει το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Ε, ήρθε ο κύριος Έριξον διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου ε, Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, που μας έδωσε μία πρώτη γνώμη. Συνέκρινε επίσης τα διάφορα ενδεχόμενα και πιθανότητες για ε, μελλοντική συμφωνία με βάση παραδείγματα ε, από τις καλύτερες συνεργασίες που έχουμε με μη κράτη-μέλη, τη Σουηδία και την Νορβηγία και βέλτιστες πρακτικές ανέφερε Προειδοποίησε όμως ότι θα υπάρχουν ε, καθυστερήσεις για τις διελεύσεις των συνόρων και, ε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης προειδοποίησε ε, να μην είναι πάρα πολύ νομικιστικές και ευρείες οι συμφωνίες και ουσιαστικά οι έμποροι είναι άνθρωποι που είναι ε, πρακτικοί και απαντούν με πρακτικό τρόπο σε πρακτικές αποφάσεις. Αυτά. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, ε, ζητήστε τις. Θα σας τις δώσω. Ωραία. Α, ο κύριος Μάρτιν. Just, just one brief... Μια σύντομη παρατήρηση μόνο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω στην ομάδα παρακολούθησης. Δεν θέλω να πω τώρα σε ε, λεπτομέρειες για τα τελωνιακά, αλλά τι είπε όμως ο κύριος, ε, υπονόησε ή υπέδειξε ως καλύτερο παράδειγμα το Σουηδικό. Αυτό λύνει το θέμα της Βορειοϊρλανδίας ή όχι. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ε, πολιτικά φορτισμένο και εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχουν οδηγίες με την Ορβηγία και τη Σουηδία Ε, αυτοί έχουν σύνορα πάρα πολύ ε, μακρά. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο το θέμα στην Βρετανία και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες σύνοριακές διελεύσεις, υποθέτω. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Τα αγαθά δεν θα περνούν τα σύνορα όπου να είναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μεθοριακός σταθμός και ε, θα έχει συμφωνηθεί. Ε, από τεχνική σκοπιά αυτό είναι δυνατό, αλλά πολιτικά εναπόκειται στη, στο Λονδίνο, στη και όπου πολλού λαμβάνονται αποφάσεις. Ωραία. Άλλο τίποτα, συνάδελφοι, προς τους εισηγητές για το θέμα των ομάδων παρακολούθησης. Όχι. Ωραία, να κλείσετε αυτό το θέμα και το επόμενο ε, αφορά το Μαρόκο. Το 19 η πορεία των διαπραγματεύσεων με το Μαρόκο όσον αφορά τι συμφωνίε σχετικά με την προσαρμογή των πρωτοκόλων για του κανόνε καταγωγή στο πλαίσιο τη Συμφωνία Σύνδεση και τη Αλληλευτική Συμφωνία. Είναι και το τελευταίο μα θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Και αποφάσισαν οι συντονιστέ μετά από το αίτημα τη κυρία Λαλόντ, τη εισηγήτρια, να ενημερωθούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το πού βρισκόμαστε στις τόσο σημαντικές αυτές διαπραγματεύσεις. 20 Φεβρουαρίου η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενημέρωσε την Επιτροπή μας για το περιεχόμενο της μελλοντική αυτής ε, συμφωνίας και ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η διαβούλευση ώστε να ικανοποιηθεί το... η απόφαση του Δεκεμβρίου του 2016 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ούτε το, η τροποποίηση του πρωτοκόλου, ούτε οι ελληνικέ συμφωνίες δεν ενημερώθηκαν από το Σώμα των Επιτρόπων, όπως γνωρίζω. Οπότε, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος αυτός είναι πολυδιάστατος. Ενδιαφέρει την ΑΦΕΤ, την ε, Επιτροπή Αλίας, και άλλοι ζήτησαν ε, να συμμετάσχουν μεν χωρίς να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους οι ευρωβουλευτές. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πατρίσια Λαλόντ που είναι η μόνιμη εισηγήτριά μας για αυτό το θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Sorry, but uh, I lost my glasses. Έχασα τα γυαλιά μου οπότε μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω, έχασα τα γυαλιά μου. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντο και τη Γενική Διεύθυνση Μάρα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να έρθουν να ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε κάποια πρόοδος από την προηγούμενη φορά που συνδυάσαμε για αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τώρα το περιεχόμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Συνεπώς, πολύ σύντομα θα μας στάσει ο φάκελος, πολύ σύντομα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου το Συμβούλιο, 16 Απριλίου που μας πέρασε, έκρινε την εντολή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελληνική Συμφωνία. Χτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είχαμε τον κύριο Σκουλ που είναι ο αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Σαχάρα και μα εξήγησε πώ βλέπει την αποστολή του και ποιοι θα είναι οι στόχοι. Επί τη ευκαιρία αυτή επαναλάβαμε ότι στηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία από τον ΟΗΕ, η αποστολή ειδικού αντιπροσώπου, ειδικού απεσταλμένου, συγγνώμη. Μπορεί να μην συνδέεται άμεσα με τι αρμοδιότητε τη δική μα ε, επιτροπή, Η ειρηνευτική διαδικασία όμω αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφεται και η δική μας δράση. Οπότε είναι ζωτική σημασία στο δικό μας έργο εδώ να γράφεται ακριβώς στα πλαίσια και της στήριξης του ειδικού αυτού απεσταλμένου. Μας εξέπληξε η πραγματική επιθυμία, η έντονη βούληση να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε ξανασυναντηθεί εδώ με την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Τώρα ε, θέλουμε αυτή η νέα ανταλλαγή απόψεων να μας επιτρέψει πρώτο να καταλάβουμε πόσο έχει προχωρήσει η υπόθεση, πόσο έχει προσαρμοστεί δηλαδή η Συμφωνία Σύνδεσης και να μιλήσουμε για την επαναδιαπραγμάτευση της αλλιευτικής συμφωνίας σχετικά με την οποία το Φεβρουάριο που μας πέρασε ε, εξέδωσε απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλουμε πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τη διάρθρωση των δύο αυτών ζητημάτων και επίσης να ακούσουμε τι προσαρμογή στην Ελευτική Συμφωνία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα ζητήματα που με απασχολούν είναι τα εξή και από εκεί και πέρα θα επιτρέψω στους συναδέρφους να συμπληρώσουν τι ερωτήσει. Μπορείτε να μα πείτε με λεπτομέρεια πού βρίσκεται η διαδικασία για την Συμφωνία σύνδεση και να μα πείτε πότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να περιμένει να του υποβληθεί η υπόθεση αυτή. Υπήρχε μια προθεσμία, ισχύει πάντα. Υπάρχει και νέα εξέταση, προβληματισμός που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας από βράση επιτροπής δηλαδή για στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη διαβούλευση. Και τέλος, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την αλληλευτική συμφωνία, το χρονοδιάγραμμα της νέας αυτής συμφωνία και τη σχέση της αλληλευτικής συμφωνίας με την συμφωνία σύνδεσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Λυπάμαι που χάσατε τα γυαλιά σας, ελπίζω να τα βρείτε σύντομα. Αλλιώς θα πρέπει να αγοράσετε. Λοιπόν, οι πολιτικές ομάδες. Η Μαρία Ρένα πρώτα, εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ε, ελπίζω να είναι έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πατρίσια. Και εγώ συμμετείχα στην ακρόαση του ειδικού απεσταλμένου χτες. Όντως, το έργο των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να στηριχτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ίδιος περιμένει πολλά από μας. Εδώ στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, δεν βλέπω συναδέρφους εδώ ούτε από την Επιτροπή Γεωργίας ούτε από την Επιτροπή Αλίας, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε περισσότερο οριζόντια να συνεργαζόμαστε για αυτά τα θέματα μεταξύ μας, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στόχος μας είναι να υπάρχει σταθερότητα στις σχέσεις μας με το Μαρόκο και κυρίως τις εμπορικές μας σχέσεις με το Μαρόκο. Και όταν ε, λέμε σταθερότητα, αυτό είναι σημαντικό για τους επενδυτές επίσης. Να γνωρίζουν δηλαδή ποιο είναι το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν, ώστε να μπορούν να επενδύσουν στο Μαρόκο. Και το Μαρόκο τη χρειάζεται αυτή τη σταθερή σχέση επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθερή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει νομική σταθερότητα. Δουλεύουμε όχι στα πλαίσια μιας παραδοσιακής σχέσης με το Μαρόκο, αλλά αντιδρούμε σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει, τμήματα των οποίων θεωρήθηκαν είτε μη ικανοποιητικά ή ατελή, προκειμένου να σεβαστούμε τις, τα διεθνή πρότυπα, τις διεθνείς συμφωνίες, κυρίως για τη Δυτική Σαχάρα. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι η συνένεση για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Είτε πρόκειται για την αλληλευτική, είτε πρόκειται για την συμφωνία για τα γεωργικά. Ξέρω ότι το θέμα της συνένεσης αυτής είναι δύσκολο, γιατί τι σημαίνει ακριβώς, ποιος πρέπει να συνενέσει, πώς θα γίνουν οι διαβουλεύσεις. Ξέρω ότι σήμερα υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τις αρχές του Μαρόκου. Χρειάζεται διαφάνεια λοιπόν. Και η θέση μου είναι από τη στιγμή που αυτό το εγχείρημα της συνένεσης είναι τόσο δύσκολο, είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποφάνθηκε για τη συνένεση αυτή άρα να ακούσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει να επιτυχάνεται η συνένεση αυτή από τις ε, διαπραγματευόμενες πλευρές. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε τη θέση του δικαστηρίου και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να θέσουμε το θέμα της ψηφοφορίας επί των συμφωνιών αυτών, να έχουμε απάντηση από το δικαστήριο κατά πόσο οι διαδικασίες διαβούλευσης που έλαβαν χώρα από το Μαρόκο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφονται στην λογική αυτή της συνένεσης που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έχω μία ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα. Λίγη στις 14 Ιουλίου η Αλληλευτική Συμφωνία. Σήμερα είμαστε μέσα Μαΐου. Αν θέλουμε όλη αυτή η δουλειά να γίνει μέσα στην προθεσμία που έχουμε, δεν πρέπει να την κάνουμε και κλειμένο των θυρών αυτή τη δουλειά. Ενώ αυτό γίνεται σήμερα. Διαπραγματεύονται η Επιτροπή με το Μαρόκο και εμεί δεν συμμετέχουμε καθόλου. Αν θέλουμε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετηθεί πριν από τις 14 Ιουλίου, όπως θα έπρεπε, είναι αναγκαίο να πάμε πιο γρήγορα και να έχουμε και περισσότερη διαφάνεια και να μην ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετείται χωρίς να έχει στη διάθεσή του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να τοποθετηθεί ακριβώς ε, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τέλος, άκουσα κάποιους συναδέρφους να λένε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θέτει σε κίνδυνο τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Απαντάω σε αυτούς τους συναδέρφους ότι το να συμμορφώνεται κανείς με τη δικαιοσύνη δεν σημαίνει ότι θέτει σε κίνδυνο μια συμφωνία. Αντίθετα, όταν δεν συμμορφωνόμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις, τότε θέτουμε σε κίνδυνο συμφωνίες όπως αυτή που έχουμε με το Μαρόκο. Γι' αυτό ζητάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σεβαστεί τη δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να περάσουμε στο συνάδελφο Χέλμουτ Σόλτς. Έχετε το λόγο. Ε, καλώς. Νόμιζα ότι θα πρέπει να μιλήσει άλλος συνάδελφος, η πράσινη δηλαδή. Ε, ο δικός μας σκιώδης απουσιάζει. Ε, συμφωνώ με την κυρία Ρενά. Δεν μπορούμε να ψηφούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα για μας της ενωτικής αριστεράς. Υπάρχει μια σαφής δήλωση που λέγει ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, διαπραγμάτευση και συνένεση. Και συνένεση θα πρέπει ε, ε, ότι μόνο διεθνώς αναγνωρισμένες δομές θα πρέπει να συμμετέχουν, που είναι το μέτωπο πολυσάριο για το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Αυτοί τους έχουν ορίσει επίσημους αντιπροσώπους τους. Εάν δεν έχει συμφωνήσει λοιπόν το Πολυσάριο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, σήμερα θέλω μια σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί και την περασμένη φορά υπεκφυγές ακούσαμε. Πώς θα το χειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να συνεχίσει να αγνοεί ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι βεβαίως οι εμπορικές σχέσεις με το Μαρόκο και η ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο και ενδεχομένως και μια ευρύτερη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο ε, είναι σημαντικό και με το λαό των Σαχράουι. Είναι πολύ σημαντικό και για τη δική τους την ανάπτυξη. Εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και θέλω μια σαφή απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που άλλαξα τη σειρά των πολιτικών ομάδων. Τώρα η πράσινη και ο κύριος Μποχνερ που έπρεπε να μιλήσει προηγουμένως. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξανατονίσω το εξή. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εντολή την εμπορική έχει σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ε, γλωσσική έκδοση στα αγγλικά γίνεται λόγος για το, τους people of Western Sahara ενώ στα γαλλικά population, δηλαδή στη μια περίπτωση είναι λαός και στην άλλη είναι πληθυσμός. Δηλαδή, στη μία περίπτωση είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί και στην άλλη περίπτωση είναι οι άνθρωποι που κατάγονται από εκεί. Ο λαός της Δυτικής Σαχάρας που λέγονται Σαχράουι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν όταν πρόκειται για το ίδιο έγγραφο στα γαλλικά να λέει κάτι τελείως διαφορετικό από το αγγλικό. Ε, το δεύτερο ε, στο οποίο θα θέλω να αναφερθώ είναι η διαφορά ανάμεσα στη συμφωνία ε, για τα γεωργικά προϊόντα και για τα αλλιευτικά προϊόντα. Στη μία περίπτωση πρόκειται για απλή προσαρμογή ε, των κανόνων ε, καταγωγής των προϊόντων, ενώ στην, αυτό στη Γεωργία, ενώ στην Αλία γίνεται ρητή αναφορά στον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Και τέλος, για να το διευκρινίσουμε, ποιο είναι το θέμα. Οι διαπραγματεύσεις τώρα θα γίνονται αποκλειστικά στη Ραμπάτ και στις Βρυξέλλες. Μα οι άνθρωποι που είναι από τη Δυτική Σαχάρα, πώς να πάνε στη Ραμπάτ, όπου τους περιμένουν όλες αυτές οι ε, διώξεις και καταστολή. Πώς το διανοήθηκε καν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί βάση μαροκινού δικαίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να ε, μετέχει πλήρω στις διαπραγματεύσει ο λαός της Δυτικής Χάρας. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, μια συμφωνία θα πρέπει να πληρεί ε, ε, τα πρότυπα και τα αποτελέσματα και, και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλιώς είναι άκυρη. Γι' αυτό με ενόχλησε αυτό που είπατε εσείς κύριε Βίνκλερ. Ότι μιλήσατε για ένα αίτημα, μια παράκληση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Καθόλου παράκληση. δικαστική απόφαση είναι και οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κι άλλο γύρω μιλητών. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω και με τις απόψεις των συναδέλφων. Σαφώς και θέλουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με το βασίλειο του Μαρόκου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σεβαστούμε και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αυτών όλων. Και θα ήθελα να τονίσω, όπω τόνισαν και οι συνάδελφοι, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε απλώ μερικέ λεξούλες ε, στη συνθήκη. Πρέπει να αλλάξουμε και πρακτικές. Επειδή αδυνατούμε μέχρι τώρα να κάνουμε κάτι για τα αγαθά προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη από το Ισραήλ και αυτές τις ομάδες. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξασφαλίσει ότι αν όντω αλλάξει η σχέση μεταξύ ημών και του Μαρόκου για να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, θα μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη χνηλασιμότητα των προϊόντων που έρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι της Δυτικής Σαχάρας θα ωφελούνται από ε, τα προϊόντα αυτά και τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Και επίσης ήθελα να ενισχύσω αυτό που είπε ο Χέλμουντ Σόλτς. Θέλουμε να έχουμε σαφείς ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιους έχουν διαβουλευτεί μέχρι τώρα στη διαδικασία, μια σαφή δήλωση ε, ποιοι είναι οι συνομιλητές τους και ποιοι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρτσελέση έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω για την ανάγκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τους νόμους της και να σέβεται κυρίως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για μένα είναι θέμα και αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοπιστίας. Και πραγματικά ε, τι αξιοπιστία δίνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπω ε, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ερωτήσει που έχουμε θέσει επανειλημμένω και ακόμα δεν έχουμε λάβει σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δύο φορέ μας λέει σαφώς ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι συγκατάθεση του λαού της ε, Δυτικής Σαχάρας. Όχι μόνο διαβούλευση, αλλά συγκατάθεση. Και αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μια διαδικασία διαβούλευσης που γίνεται μεταξύ Βρυξελών και Ραμπάτ. Ε, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί από του κατοίκου τη Δυτικής Σαχάρα και του εκπροσώπους δεν μπορούν να, καν να πάνε στο ραμπάτ και όταν πηγαίνουν δεν μπορούν να μιλήσουν καν ανοιχτά για τη διαδικασία τη αυτοδιάθεση, το οποίο αναγνωρίζεται και διεθνώ. Επομένω, θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια διαβούλευση ανοιχτή και διάφανη και ταυτόχρονα να λάβει και αυτή τη συγκατάθεση. Πώ σκοπεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρει να έχει τη συγκατάθεση του λαού τη Δυτικής Σαχάρα. Δεύτερον, και αυτό έχει σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Αλευτική Συμφωνία. Διότι ε, το δικαστήριο λέει στην παράγραφο 76 ότι το Μαρόκο αρνείται να αναγνωριστεί με άλλο τρόπο, δηλαδή ως κυρίαρχη δύναμη ε, στη Δυτική Σαχάρα. Επομένως, ουσιαστικά το δικαστήριο λέει ότι δεν μπορεί να είναι κυρίαρχη δύναμη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Ε, και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Επομένω, τι ε, μπορείτε να κάνετε, πώ μπορείτε να διαπραγματευτείτε με το Μαρόκο όταν δεν έχει αυτό την κυριαρχία και δεν έχει νομική σχέση ε, για τη Δυτική Σαχάρα. Και επομένω αυτό είναι και η βάση οποιασδήποτε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου και σε αυτή την περίπτωση και Δυτική Σαχάρα. Και όπως είπε και η Μαρία Ρενά, θα πρέπει να υπάρχει και μια γνωμοδότηση του δικαστηρίου για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφανθεί εάν δεν έχει πρώτον τη σαφήνεια ότι ε, σωστά κάνουμε αυτά που κάνουμε. Διότι υπάρχουν ε, χρόνια έλλειψη ασφάλεια δικαίου. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή οι αλληλείς από τη Γαλλική, από την Ανδαλουσία που θα πάνε να ψαρέψουν εκεί και το 80% είναι από τα ψάρια της Δυτικής Σαχάρας, αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε νομικό κενό. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίωση. Ποιο θα πληρώσει γι' αυτό, ποιο ε, θα πληρώσει γι' αυτή την ευθύνη. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά πρόκειται για ένα θέμα αξιοπιστία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σαφώς σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μινέρ για να ολοκληρώσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προηγουμένω συζητούσαμε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είναι σαφή. Η αλληλευτική συμφωνία ε, με το Μαρόκο δεν ισχύει για τη Δυτική Σαχάρα εκτό αν έχει συνενέσει ρητά ο εκεί πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αυτή τη συνένεση ούτε προσπαθεί να την αποσπάσει ή να την αποκτήσει. Ε, συζητάει με τον κατακτητή, με εκείνου που έχουν ε, υποκατοχή την επικράτεια και όχι με το λαό των κατεχομένων και με την ενευτική αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προτίθεται να ακολουθήσει το γράμμα του νόμου και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να ζητήσει ρητά τη συνένεση και οι χώρες ε, ΕΖΕΣ και ε, το, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συμφωνίες τέτοιες με το Μαρόκο που εξηρεί τη Δυτική Σαχάρα. αλλά αυτό μπορεί να γίνει. Και υπάρχει και άλλη ομάδα εκτός από τους Σαχράουι που υφίσταται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στην οροσυρά του Ριφ. Τι γίνεται εκεί λοιπόν με τον λαό αυτό και ε, στην αλλιευτική συμφωνία, στη γεωργική συμφωνία και στην ε, υπόλοιπη συνεργασία που έχουμε με το Μαρόκο. Λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο της διαφθοράς και τα δικαιώματα του λαού της οροσυράς Ριφ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές ερωτήσεις και θέλουμε να έχουμε απαντήσεις παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κριστιαν Ραμπό ονομάζομαι και είμαι τμήματάρχης στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ που ασχολείται με την Ελληνική Συμφωνία. Οπότε θα απαντήσω σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελληνική Συμφωνία και είμαι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Μαρόκο. Μια επενθύμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά εργάζεται, ακόμα και αν στις 17 Απριλίου άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, εργαζόμαστε καθημερινά για να βρούμε λύση που να τηρεί βέβαια την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπενθυμίζω ότι η απόφαση αυτή στα συμπεράσματα λέει ότι η ελευτική συμφωνία είναι νόμιμη, αλλά μόνο στα ύδατα τα οποία είναι δικαιοδοσία της χώρας του Μαρόκου. Κάτι το οποίο βέβαια αποκλείει τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Συνεπώς, τι κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση η οποία να επιτρέπει στο πνεύμα αλλά και στο γράμμα της δικαστικής αυτής απόφασης να βρούμε μία λύση η οποία να επιτρέπει να συνεχίσουμε τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, σήμερα βρισκόμαστε σε μία κατάσταση νομικής ε, αβεβαιότητας με σημαντικές οικονομικές ε, συνέπειες, είτε πρόκειται για τους Ευρωπαίους που δρούν στα ύδατα αυτά παραδοσιακά, είτε πρόκειται για τον ε, κόσμο που ζει στα παράκτια. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια λύση. Αυτή η λύση ε, πάει λίγο σημειωτών, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε μια επιλογή. Τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Εργαλεία μέσα, τα οποία να είναι του ίδιου νομικού χαρακτήρα. Πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες. Γιατί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι αντίθετα με αυτά που λέει η ε, συμφωνία Γεωργίας που είναι η Συμφωνία Σύνδεση και τα πρωτοκόλλα 1 και 4, αυτά που ισχύουν και που θεωρεί το δικαστήριο ότι ισχύουν αλλά μόνο σε ένα τμήμα των υδάτων, είναι μια παλιά συμφωνία. Στο μεταξύ υπήρξε νέα θήκη, η Λισαβόνα, άρα δεν πρόκειται πια για συμφωνία ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μαρόκου, πρόκειται Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκο. Δεύτερον, η κοινή ληφτική πολιτική μεταρρυθμίστηκε το 2013. Μετά δηλαδή από την συμφωνία που ισχύει τώρα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο η συμφωνία αυτή με το Μαρόκο να ευθυγραμμιστεί στις νέες αρχές, στους νέους στόχους που έχουμε στον βασικό μας κανονισμό και που έχουν στόχο ε, να ε, επανακτηθεί μια βιώσιμη αλία. Και όλα αυτά περνάνε ε, μέσα από την πρόσβαση των Ευρωπαίων στα αποθέματα, πλονάσματα μάλλον, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αλία. Αυτό σημαίνει επίσης να μην υπάρχει διάκριση σε βάρος ε, του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλων χωρών και δεν πρόκειται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο που δρούν στα ύδατα αυτά, δρούν και πολλοί άλλοι. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να θέλουμε μια νέα ε, βιώσιμη αλληλευτική συμφωνία. Ο σημερινός μας στόχος είναι να δούμε, πρέπει αναλογικά να προχωρήσουμε, αναλογικά δηλαδή με το σύστημα που παρακολουθεί τα γεωργικά ζητήματα στη Συμφωνία Σύνδεσης. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια συμφωνία που να συμπληρώνεται από ανταλλαγή επιστολών ίσως και από ένα πρωτόκολλο. Δεν θα μιλήσω για το πρωτόκολλο, αλλά και εδώ δεν πρόκειται για την απόφαση του δικαστηρίου που μας αναγκάζει στην ανανέωση του πρωτοκόλλου, απλώς το σημερινό πρωτόκολλο εκπνέει στις 14 Ιουλίου φέτος. Συνεπώς, οι εργασίες μας για την αξιολόγηση, την προετοιμασία και για την εντολή που έδωσε το Συμβούλιο στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί το νέο πρωτόκολλο, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτά τα τρία αντικείμενα πρέπει να συζητηθούν με το Μαρόκο για να βρούμε μια λύση. Τώρα επί της αρχής υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία εδώ. Το πρώτο είναι ο ορισμός του πεδίου εφαρμογή βέβαια. Το πεδίο εφαρμογή καλύπτει τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας χωρίς να αναγνωρίζει εφόσον το λέει το δικαστήριο την αρχή της κυριαρχίας ή της δικαιοδοσίας του Μαρόκου στα ύδατα αυτά. Άρα λοιπόν η δυσκολία εδώ είναι να βρούμε ε, μια λύση η οποία να είναι νομικά δεσμευτική, αλλά και από την άλλη να μην είναι σε αντίφαση με την απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, τα ωφέλη στον πληθυσμό από τα κέρδη. Εδώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την ορολογία ε, της εντολής του Συμβουλίου. Εδώ γνωρίζετε ότι αντίθετα από ό,τι ισχύει στη Συμφωνία Σύνδεσης, η Αλληλευτική Συμφωνία προβλέπει κονδύλιο το οποίο αποτελείται από τρία στοιχεία. Πληρώνουμε για την πρόσβαση στα ύδατα, οι εφοπλιστές πληρώνουν για να δρούν στα ύδατα αυτά και έχουμε επίση και στήριξη στην ε, τομεακή πολιτική, την ελευτική δηλαδή. Πρόκειται για τρία στοιχεία πρόθεσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι στα τρία αυτά στοιχεία, στις τρεις αυτές συνιστώσεις, να γίνεται κατανομή στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό επιτόπου. Και το άλλο είναι ότι όλες οι διαδικασίες τις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, κάτι που δεν υπάρχει στη σημερινή συμφωνία, αλλά το προτείνουμε για την επόμενη, είναι να υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιείται από τη στιγμή που θα υπάρξει αποτέλεσμα. Τέλος, όσον αφορά τα ωφέλη του πληθυσμού, στο σημερινό πρωτόκολλο υπάρχει αυτή η στήριξη στον κλάδο που την παρακολουθεί μια μεικτή επιτροπή, η οποία κάθε χρόνο ο αξιολογεί, εκτιμάει βάση του αρχικού προγραμματισμού που έχει υποβάλει το Μαρόκο και εγκρίνει η μεικτή επιτροπή άρα και Ευρωπαϊκή Ένωση, μας επιτρέπει λοιπόν να επαληθεύουμε ότι όλα τα στοιχεία, όλες οι παράμετροι που έχουν προγραμματιστεί, τηρούνται κιόλα. Και σας καλώ να διαβάσετε την αξιολόγηση ex post και ex ante που έγινε ε, για τη συμφωνία με το Μαρόκο, τη σημερινή, από την οποία και εμπνεύστηκε εξάλλου το δικαστήριο για να πει ότι το μεγαλύτερο μέρος, γιατί πρόκειται πάνω από 65% της στήριξης του κλάδου, χρησιμοποιήθηκε για τις περιοχές του Νότου, είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί το Μαρόκο. Τώρα, για τη συνέχεια σας είπα ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να βρούμε λύση και για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και για τις διάφορες παραμέτρους που σας περιέγραψα. Uh, very... Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά. Uh, uh on the commission side... Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζω τον κύριο Τερόντε Πίνη και του δίνομαι στο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να σας ενημερώσουμε για την ε, τροποποίηση της συμφωνίας ε, σύνδεσης. Θα θυμάστε ότι υπήρξε μια αλληλογραφία ε, που ολοκληρώθηκε τέλη Ιανουαρίου και αυτή είναι η μορφή που θα λάβει η συμφωνία. Και τα βασικά ε, στοιχεία είναι τα εξής. Τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα θα την χάνουν των ιδίων προτιμήσεων όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του Μαρόκου. Οι κανόνες καταγωγής της Συμφωνίας Σύνδεσης θα ισχύουν εκεί με τις απαραίτητες ε, προσαρμογές και για τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης αυτής ε, με τη συμφωνία ΘΕΑ διεξάγεται από τις μαροκινές αρχές. Και όλα αυτά με την επιφύλαξη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο, των θέσεων των μερών για το ε, καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας εκφράζεται και η υποστήριξη για την ευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για να λυθεί η σύγκρουση για τη Δυτική Σαχάρα. Από την περασμένη σας συνεδρίαση οι εργασίε επικεντρώθηκαν στην οριστικοποίηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο, καθώς επίσης και σε μια έκθεση για ε, τα ευεργετήματα της Συμφωνίας για τον πληθυσμό της Δυτική Σαχάρα, και υπήρξαν και ανταλλαγέ απόψεων και διαβούλευση με ενδιαφερομένου από τη Δυτική Σαχάρα. Όλα αυτά έχουν τώρα ολοκληρωθεί σε επίπεδο τεχνικών ε, υπηρεσιακών παραγόντων και το επόμενο βήμα είναι να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η πρόταση αυτή και να ε, υπάρξει μια πρόταση στο Συμβούλιο αφενός για την υπογραφή ε, της συμφωνίας αυτής και αφετέρου για τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επισυναυθούν στην έκθεση. Όλα αυτά αναμένεται να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες, πολύ λίγες εβδομάδες. Και το θέμα που σας παρουσίασε ο συνάδελφος Γαμπό από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ είναι διαφορετικό από την Αλευτική Συμφωνία. Βέβαια, αφού πρόκειται για την ίδια χώρα, υπάρχουν κάθε... Προφανώς, ε, προφανές ότι υπάρχουν ε, ομοιότητες και συμπτώσεις για τη Δυτική Σαχάρα. Αυτά ήθελα να πω εγώ τα διαδικαστικά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αν έχετε ερωτήσει να απαντήσω ευχαρίστως πριν δώσουμε το λόγο στους ε, βουλευτές για ερωτήσεις, να μας πει η φρονεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο κύριος Νίκολας Μπούλτε, αν το λέω σωστά, σας δίνω μέσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμείς ουσιαστικά ε, συμμετείχαμε ε, στο σκέλος που αφορά τις διαβουλεύσεις. Το people concerned στα αγγλικά, ε, population concerned, ενδιαφερόμενος πληθυσμός στα γαλλικά, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων λοιπόν για τη Γεωργική Συμφωνία. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, είναι πλάκιμεν πάντα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικά για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε έγιναν αυτές οι διαβουλεύσεις και το αποτέλεσμα τους θα το δείτε στην έκθεση, τη συνοδευτική των εγγράφων που θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας αποκαλύψω το περιεχόμενο. Απλώς καταβάλαμε μια προσπάθεια με τον εξής στόχο. Να καλύψουμε όσο γίνεται ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων και σε τεχνικό επίπεδο αφού το θέμα της Γεωργικής Συμφωνίας είναι πάρα πολύ τεχνικό και εμπορικό ενώ για το πιο πολιτικό θέμα επίσης είχαμε τη μέρημνα και το μέλημα να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερο κοινωνία των πολιτών. Ε, ε, σε αυτά τα τρία λοιπόν σταθήκαμε. Έγιναν διαβουλεύσεις από τις μαροκινές αρχές με την τοπική κοινωνία, ε, την ε, τοπική αυτοδιοίκηση που εκπροσωπεί την κοινωνία. Αυτό έγινε ε, στο βαθμό του δυνατού για να καλύπτεται όσο γίνεται ο λόγο πληθυσμός και η κοινωνία των πολιτών αλλά και πολιτικοί φορείς όπως το μέτωπο Πολυσάριο ως φυσικός ε, εταίρος συμμετέχουν στην νευτική διαδικασία από την Αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματικά φροντίσαμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερους ε, ε, φορείς και ενδιαφερομένους, ιονί ενδιαφερομένους από την τροποποίηση, για την τροποποίηση αυτή. Ορισμένε από τις ε, οργανώσεις τι οποίε αποταθήκαμε δεν θέλησαν να απαντήσουν στην πρόσκλησή μας, τουλάχιστον προς στιγμή. Παραμένει ε, ανοιχτή η πρόσκληση και πάντα αυτό είναι το μέλημά μας. Όσο γίνεται περισσότεροι να συμμετέχουν. Είμαστε όσο γίνεται πιο εξαντλητικοί στην προσέγγιση μας. Έχοντας πάντα υπόψη μας ότι η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω νέο γύνορο επερωτήσεων. Να ξαναπεράσω λοιπόν στις πολιτικές ομάδες η Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για τις πληροφορίες και πράγματι έχουμε μια συμφωνία σύνδεσης και έχουμε και μια λευτική συμφωνία. Τολμώ δε να πω ότι κανονικά η Ελευτική Συμφωνία δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και αφορά αποκλειστικά την, την ε, Επιτροπή Αλληλείας, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία μα εμπλέκουν. Την απόφαση του δικαστηριού που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και συνέπεια για την απάντηση που θα δώσουμε και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα πιο οριζόντια και να μην το δούμε σε κάθε Επιτροπή ξεχωριστά. Έχω αρκετές ερωτήσεις για αυτά τα οποία μας απαντήσατε και όσον αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης και όσον αφορά την Ελληνική Συμφωνία. Πρώτον, αποφασίστηκε σαφώς από την Επιτροπή και από τις ε, αρχές του Μαρόκου να απαντήσουν στο ερώτημα του δικαστηρίου λέγοντας ότι ε, πράγματι το δικαστήριο θεωρεί ότι οι συμφωνίες είναι νόμιμες και αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο, αλλά είναι νόμιμες υπό κάποιες προϋποθέσεις. Και όσον αφορά τη Γεωργική Συμφωνία ή τη Συμφωνία Σύνδεσης, εάν θεωρείτε ότι η Δυτική Σαχάρα είναι τμήμα των συμφωνιών και αυτό αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποκλείσει τη Δυτική Σαχάρα, θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η υπόθεση, αλλά δεν χρησιμοποιείται αυτή η υπόθεση και λέμε ότι θα ε, εργαστούμε και με την περιοχή της Δυτικής Χάρας και τις άλλες περιοχές της Δυτικής Σαχάρας για την Αλία ε, το 90% του ε, καρπού της αλίας ούτως ή άλλως είναι από την ε, περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Αν θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι η αλία είναι νόμιμη, είναι μόνο ειναι νομη ειναι μονο νομη κατα 10%. Και λυπάμαι που σας το λέω κύριε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, την επομένη της υπογραφής του πρωτοκόλου, οι αρχές του Μαρόκου με πάσα διαφάνεια σας έδωσαν τους χάρτες τις περιοχές τις οποίες θα δώσουν άδειε. Και σε αυτούς τους χάρτες υπήρχαν και τα ε, χωρικά ύδατα της Σαχάρας. Το ξέρατε λοιπόν, δεν ήταν κάτι το οποίο αγνοούσατε, αλλά ως μη γενόμενο ε, υπήρχε απόφαση του δικαστηρίου και συνεχίζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο ε, και δεν ακούμε τι. Δεν είχαμε όμως και απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα έχουμε απόφαση του δικαστηρίου που λέει φτάνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Επομένω πρέπει να συμμορφωθούμε. Και αυτό είναι ο φόβο που έχω εγώ ω Ευρωβουλευτή. Εχθέ το γνωρίζατε, αλλά ε, το αγνοούσατε. Και θα ήθελα τουλάχιστον σήμερα αυτό που θα διαπραγματευτείτε να σέβεται αυτό το οποίο ζητάει το δικαστήριο. Και γι' αυτό ακριβώ και θεωρώ ότι ο καλύτερο τρόπο να γνωρίζουμε αν ε, γίνεται σεβαστό αυτό που ζητάει το δικαστήριο είναι να ρωτήσουμε το δικαστήριο εάν υπάρχει συμμόρφωση με αυτό που μα ζήτησε. Είναι μια νομική διαδικασία αυτή. Δεν ε, θέλω να επισέλθω σε μια πολιτική διαδικασία. Η πολιτική διαδικασία του καθεστώτος ε, της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι έχουμε αποφασίσει ότι θα γίνει υπό τη σκέπη του ΟΗΕ. Επομένω, δεν θα αποφασίσουμε εμεί για τη Δυτική Σαχάρα σε μια λευτική συμφωνία, με μια συμφωνία ε, σύνδεση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν υπό τη σκέπη του ΟΗΕ. Πρέπει να έχουμε όμω κάτι το οποίο να συμμορφώνεται τουλάχιστον σε αυτό που μα λέει το δικαστήριο. Όταν λοιπόν μα λέτε ότι έχετε προβλήψει μια ρήτρα αναθεώρηση. εγώ ανησυχώ από τη ρήτρα αναθεώρηση θα συμμορφωθούμε ε, στα όσα ζητά το δικαστήριο. Εγώ ζητώ η συμμόρφωση να γίνει τώρα και όχι μέσω μιας ρήτρας αναθεώρησης. Πώς λοιπόν θα υπάρξει ε, η συγκατάθεση στην Ελευτική Συμφωνία, διότι από ό,τι άκουσα υπάρχει ένα σύστημα ξεχωριστών θεμάτων για την Ελευτική Συμφωνία, αλλά όσον αφορά τη συγκατάθεση ε, θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα τι θα μας εγγύθει ότι οι διαβουλεύσεις οι οποίες είναι εξελέξει αυτή τη στιγμή θα μεταφραστούν σε πραγματική συγκατάθεση των λαών που ζουν αυτή τη στιγμή στη Δυτική Σαχάρα και για ε, των οποίων θα χρησιμοποιούνται τα χωρικά ύδατα. Το αυτό ισχύει και για την ε, Γεωργική Συμφωνία. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει δυνατότητα να προβλέψουμε, γιατί μου λένε ότι είναι κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί να υπάρχει μια προσωρινή ισχύ ε, χωρίς να υπάρχει έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ κακό μήνυμα να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα πράγματα χωρίς να υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο έχετε στα χαρτιά της διαπραγμάτευσης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μαρόκου αυτή τη στιγμή. Προβλέπετε δηλαδή να μην περάσετε από τη διαδικασία κύρωσης. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και το προβλέπετε αυτό. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μασιλές έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να είμαι ειλικρινής ε, μαζί σας. Έχω πέσει από τα σύννεφα με την ε, πρώτη απάντηση που άκουσα. Ήδη σήμερα το πρωί δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά που ρωτήσαμε. Για την συνένεση, για παράδειγμα, τη συγκατάθεση. Δεν πήραμε καμιά απάντηση. Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις που να βασίζονται σε νομικά στοιχεία για αυτή την μεικτή επιτροπή. Επίσης, δεν ακούσαμε Θέλουμε απαντήσεις και οφείλεται απαντήσεις στους ευρωβουλευτές. Έτσι είναι λογικό σε μια τέτοια συζήτηση να έχουμε απαντήσεις. Επίσης, με σόκαρε και η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ορολογία της, γιατί έχουμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πρέπει να τηρήσουμε και αναφέρεται στο λαό της Δυτικής Σαχάρας. Σήμερα το πρωί άκουσα για πληθυσμό που ζει στα παράκτια, ενδιαφερόμενο πληθυσμό, ε, τοπικό πληθυσμό. Δεν άκουσα καμιά φορά από εσά να μιλάτε για τον λαό τη Δυτική Σαχάρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί εδώ και να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του. Και όταν επιπλέον λέτε ότι αναγνωρίζετε πως δεν υπάρχει κυριαρχία του Μαρόκο στη Δυτική Σαχάρα και μετά μιλάτε για τις περιοχές του Νότου, ή λάθος είναι, ή ακόμα χειρότερα επίτηδες. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που λέει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το είπε σαφώ και ο άλλο εκπρόσωπος τη Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα διακριτό έδαφο. και χωρισμένο. Είναι σαν να λέμε για την Κρυμαία ότι είναι ρωσικά εδάφη, έτσι. Το ίδιο κάνουμε και εδώ τώρα για τη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώ. Ωραία. Δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε απαντήσει. Αν δεν έχουμε απαντήσει, τότε θα ήθελα η ΙΝΤΑ, η Επιτροπή μα, να στείλει επιστολή σαφή επιστολή με την οποία να ζητάει πολλά διάφορα. Παράδειγμα, για την ανταλλαγή επιστολών. Με τι νομική βάση γίνεται αυτή η ανταλλαγή επιστολών. Έπειτα θέλω να ξέρω αυτή η μεικτή επιτροπή. Ποια είναι η σύνθεσή τη, ποια είναι η νομική τη βάση. Είναι πράγματα που μερικές φορές δύσκολα καταλαβαίνουμε ευρωβουλευτές που έχουμε εκλεγεί, αλλά θα έπρεπε να καταλάβουμε την δικαστική απόφαση και αυτή τη συγκατάθεση πώς θα την αποκτήσετε. Θέλουμε μια απάντηση σε αυτό. Λέτε ότι διαβρύθηκε η διαβούλευση. Μιλάτε για διαβούλευση, έτσι δεν μιλάτε για συγκατάθεση. Με... Να ξέρετε όμως ότι 89 ε, οργανώσεις από τη Δική Σαχάρα δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν. Γιατί ακριβώς δεν σέβεστε αυτό το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Θέλω λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις με διαφάνεια και να δείξετε κάποιο σεβασμό στους ευρωβουλευτές και στην κοινοβουλευτική αυτή επιτροπή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριο Σόλτ είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος, ότι θέλουμε απαντήσεις και δεν τις πήραμε σήμερα. Συγκεκριμένα όμως, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης διαβουλευτήκατε με το μέτωπο Παλισσάριο που είναι ο, μόνιμος, ο, ο μόνος νόμος εκπρόσωπος του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Λέτε δεν έρχονται, τους καλέσαμε, δεν συμμετέχουν, άλλοι δεν συμμετέχουν. Άλλοι. Ναι, πρέπει όμως να υπάρχει ε, μία σαφής απάντηση από αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται, πρέπει να διαβουλευτείτε μαζί τους προκειμένου να πετύχετε τη συγκατάθεσή τους πρέπει να σας δώσουν τη συγκατάθεση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του λαού αυτού. Αλλιώς πρέπει να συνεχίσετε ή να προσαρμόσετε τη συμφωνία ανάλογα. Δεύτερον, ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων αυτών και αν δεν υπάρχει θέση από πλευρά του Συμβουλίου θα ζητήσετε νέα εντολή για ολόκληρη τη διαδικασία και για τις δύο συμφωνίες. Και συμφωνώ με την κυρία Ρένα ότι χρειάζεται μια οριζόντια προσέγγιση εδώ για τα διάφορα προβλήματα και πολύπλοκα θέματα. Ελπίζω να μπορέσετε να μας απαντήσετε, γιατί η κυρία Μογκερίνη είπε ότι οι εξωτερικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξυπηρετούν και να αποφεύγουν συγκρούσεις στις διάφορες περιοχές και όχι αντίθετα να τις εντείνουν. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς με κάλυψε και έκανε την ερώτηση που ήθελα να κάνω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αφήσω ε, τελευταία την εισηγήτρια, κυρία Μινέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για βάλτε ακουστικά. συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους και υποστηρίζω ε, αυτή την έκκληση, την επίγουσα να απαντήσετε. Και σας θυμίζω αυτό που ρώτησα εγώ για τους κατοίκους της οροσυράς του ΡΙΦ, γιατί αυτούς τους βαρβερίνους δεν πήρα απάντηση. Uh, Ωραία. Η συγκήτριά μας η κυρία Λαλόντ για να κλείσει. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Πολλά υπόθηκαν και πολύ ενδιαφέροντα. Τα ακούσαμε και χτες με τον κύριο Χαν Κόλλερ. Με τις προθεσμίες τι γίνεται θα ήθελα να ρωτήσω εγώ. Δεν μας απάντησαν. Κάτι άκουσα για τον Ιούνιο στο Κοινοβούλιο. Ισχύει αυτό. Γιατί ε, ε, τις προάλλες άκουσα ότι στο Κοινοβούλιο θα φτάσει το Σεπτέμβριο το θέμα αυτό, μετά ε, τις θερινές διακοπές. Το Ιούνιο ισχύει, δηλαδή ο κύριος Κόλλερ θέλει να κάνει την έκθεσή του το Σεπτέμβριο, να την υποβάλει για τον Οκτώβριο. Καλό θα ήταν να συμπίπτει χρονικά αυτό. πώς μπορούμε να πάρουμε εμείς μια απόφαση για τη Γεωργία και την Αλία ετεροχρονισμένη. Καλό θα ήταν να συμπίπτει με το θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά που θέλετε εσείς. Ας απαντήσετε όπως θέλετε στις ερωτήσεις αυτές που έγιναν όλες. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη. Που μιλώ πρώτος. Ε, δεν ακούσαμε τις ερωτήσεις εμείς από τη Γενική Διεύθυνση Ταξούτ, γιατί στο Συμβούλιο είχαμε ταυτόχρονα μια άλλη συνεδρίαση. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που άκουσα τώρα, όσο μπορώ, αν τις κατάλαβα. Ε, για τη νομική βάση πρώτα. Εμείς τι κάνουμε τροποποίηση της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης επαφιέμεθα στους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την παράταση της συμφωνίας με τη Δυτική Σαχάρα ή, ή για την ε, μάλλον επέκταση της συμφωνίας για να καλύπτει και τη Δυτική Σαχάρα δεν μας δίνει 100% ε, ξεκάθαρη καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι στη Συμφωνία Σύνδεσης, και αυτό είναι το κομβικό, δεν δημιουργούμε εμεί υποχρεώσεις, ούτε επιβάλλουμε στη Δυτική Σαχάρα και στο λαό ε, της και στον πληθυσμό της οτιδήποτε ε, πλεονεκτήματα τους ε, χωρούμε. Τη δυνατότητα να επωφελούνται από τις προνομιακές ρυθμίσεις, να ε, εξάγουν αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αδασμολόγητα τα προϊόντα που παράγονται στη Δυτική Σαχάρα. Και αυτό είναι αντικείμενο διαβούλευσης όπου ηγείται η υπηρεσία εξωτερικής δράση. Αυτό που ήταν σημαντικό για μας είναι να γνωρίζουμε τις απόψεις ε, εκείνων που ε, είναι κάπως αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας, αν θα τους ε, ωφελήσει ή όχι η συμφωνία. Ουσιαστικά δεν ακούσαμε καμία αντίδραση που να θεωρούν αρνητική επιβλαβή για την οικονομία τους και για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη της περιοχής. Well known, but οι λόγοι, αν υπάρχουν λόγοι η αντίδραση, είναι πολιτική, δεν είναι οικονομική. Το θέμα ε, ήταν να διαπραγματευτούμε και να οριστικοποιήσουμε μια εμπορική συμφωνία με στόχο να ε, επεκταθούν ε, αυτά τα πλεονεκτήματα και προς τη Δυτική Σαχάρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα τώρα του πληθυσμού ή του λαού, αυτό είναι θέμα ορολογίας. Η λέξη people στα αγγλικά μπορεί να μεταφραστεί στα γαλλικά είτε peuple είτε population, δηλαδή μπορεί να είναι και ο λαός και ο πληθυσμός. Και πώς ορίζεται ο λαός της Δυτικής Σαχάρας. Ποιοι είναι, είναι αυτοί που μένουν εκεί, που κανονικά ε, μπορεί να είναι ένα κριτήριο. Ως criteria of... Τι θα βάλουμε κριτήριο προέλευσης, καταγωγής, εθνοτικό, μέχρι πού θα το πάμε. Δεν είναι δυνατό αυτό. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορούν να διεξαγάγουν εκεί συστηματική διαβούλευση ή δημοψήφισμα. Δεν έχουμε ούτε την εξουσία, ούτε το κύρος, ούτε τη δυνατότητα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, ρωτήσουμε ε, όσο γίνεται περισσότερους για να πάρουμε τις απαντήσεις και να δούμε τις απόψεις τους. σε περίπτωση που προσβληθεί ε, ε, αυτό ε, που θα αποφασίσουμε, που προσφύγει κάποιος, κληθεί να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνοι που θα πρέπει να δεχθούν, να εγκρίνουν τη συμφωνία, πρέπει να απαντήσουν στο εξή ερώτημα. Ο πληθυσμό στη Δυτική Σαχάρα θα είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα εάν του δοθούν αυτέ οι προτιμήσει. Και αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό τώρα ή να αναβληθεί και να περιμένουμε άλλα πόσα χρόνια ε, διατηρώντας αυτή την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Απαντώ στις άλλες ερωτήσεις. Αν έχετε ακόμα ερωτήσεις, ε, μη διστάσετε, θα σας απαντήσουμε βεβαίως. Πολλά από αυτά τα στοιχεία που ρωτάτε θα τα βρείτε στην έκθεση για τα ωφέλη και για τη διαβούλευση. Μου καθυστέρησε λίγο, αλλά είναι εκτενέστατη και ε, πολύ περιστατωμένη. Καλά, δεν είναι και πυρηνική φυσική, αλλά θα είναι χρήσιμη. Είναι... Ε, τώρα το θέμα του χρονοδιαγράμματος. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει εκτός απρόπτου τον Ιούνιο ε, ε, την πρόταση αυτή. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος ε, για τη μετάφραση των κειμένων και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θέμα εβδομάδων. Τώρα δεν μπορώ να σας δώσω την ακριβή ημερομηνία γιατί εξαρτάται από αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Το αργότερο μέσα Ιουνίου θα έχει εγκριθεί η πρόταση και δημοσιευθεί. Τώρα, για το πώς και με ποιον τρόπο θα πρέπει να χειριστούμε τα θέματα της αλληλευτικής συμφωνίας και της τροποποίησης ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης είναι δικό σας θέμα. Σε ό,τι αφορά την προσωρινή εφαρμογή, τα μια ερώτηση σχετικά. Όπως γνωρίζετε, η Επίτροπος Μάνστρομ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ ενώπιόν σας ε, τοποθετήθηκαν για την προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν έχει την πρόθεση να προτείνει ε, προσωρινή ε, εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών εκτός ε, κάποιων εξαιρέσεων πριν δώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία. Αυτό για τη Συμφωνία Σύνδεσης, που είναι εμπορική συμφωνία μπορεί να είναι διαφορετικές οι περιστάσεις για άλλες συμφωνίες, όπου μπορεί να υπάρχουν προθεσμίες. Αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές και θα το αποφασίσουν. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτές οι προθεσμίες ή η εκπνοή υφιστάμενων ε, συμφωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Η Γενική Διευθύνση Μάρα έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τα θέματα της ελλείας, Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φερνάντο, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούν και τις δύο συμφωνίες. Να επανέλθουμε λίγο στην αλληλεία και τα θέματα τα οποία θίξατε. Είπα στην εισαγωγή μου ότι το δικαστήριο είχε πει ότι το ε, ε, η συμφωνία είναι νόμιμη, αλλά ισχύει για συγκεκριμένη δικαιοδοσία, αποκλείοντα λοιπόν τι κείμενε περιοχέ. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο θα δεχόντουν να ε, αποφασίσουμε εμείς για το καθεστώς αυτών των υδάτων που είναι ε, στο μεγαλύτερο του βαθμό χωρικά κατά της Δυτικής Σαχάρας και ε, γι' αυτό και ανέφερα την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει μια νέα συμφωνία. Και εμεί έχουμε διεθνεί υποχρεώσει, αλλά και κοινοτικέ υποχρεώσει, κοινή αλληλευτική πολιτική, η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική επί του θέματο, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη, βιώσιμη αλληλεία βάσει των όσων προβλέπονται. Επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας μας. Αυτά τα ύδατα δεν μπορούν να είναι και, κενά. Να μην, ε, θα πρέπει λοιπόν κάπως να λαμβάνονται υπόψη και οι δραστηριότητε που γίνονται εκεί. Και να πω ότι υπάρχουν 30 χρόνια, ε, μάλλον έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που έχουμε συμφωνία για τα ύδατα αυτά και είναι ένα από τα αποθέματα αλλιευμάτων που τυχάνουν τις καλύτερες δυνατή διαχείριση ε, στα αφρικανικά ύδατα. Τώρα, όσον αφορά τα ωφέλη και τις υποχρεώσεις έχουμε την πρόθεση όσον αφορά την αλληλευτική συμφωνία να κάνουμε ό,τι ακριβώς ε, είπε και ο συνάδελφος Νικολά. Δηλαδή, να διαβουλευτούμε με τα συμβαλόμενα μέρη ε, βάσει της ίδιας διαδικασίας. Ως προς την ουσία. Θα πρέπει να γνωρίζετε και σας το εξήγησα αυτό ότι ήδη αξιολογήθηκε ένα τμήμα των ε, ωφελιών ε, του πρωτοκόλλου που έχουμε αυτή τη στιγμή ενισχύει, μέσω και της ε, εκ των υστέρων αξιολόγησης, αλλά έγινε και εκ των προτέρων αξιολόγηση. Επειδή λοιπόν η Επιτροπή σας δεν είναι ίσως εξοικειωμένη με τα θέματα λίας, σε μια συμφωνία λίας, όπως σας είπα, υπάρχουν διάφορα συστατικά στοιχεία. Στην περίπτωση του Μαρόκου σας έδωσα κάποια στοιχεία. Η συμφωνία είναι 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 16 εκατομμύρια είναι τα δικαιώματα πρόσβασης στα ε, ύδατα και πόρους και 14 ε, εκατομμύρια είναι τομεακή στήριξη και κάθε χρόνο προστίθενται βάσει των αποφάσεων 8 ε, ή 10 εκατομμύρια ευρώ που δίνουν οι εφοπλιστές. Αυτά λοιπόν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, η Μικτή Επιτροπή, εδώ να απαντήσω και ότι η νομική βάση της Μικτής Επιτροπής βρίσκεται στην συμφωνία και μάλιστα έχει τελειοποιηθεί στο πρωτόκολλο, δηλαδή καθορίζουμε την αποστολή, τη, την αποστολή της, τη λειτουργία της και την εκπροσώπηση των μελών της Μικτής Επιτροπής. Και η Μικτή Επιτροπή υπενθυμίζω ότι είναι μεταξύ των αρχών του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ένωσης. Άρα, σήμερα τα 16 εκατομμύρια ευρώ Συγγνώμη, τα 14 εκατομμύρια που αφορούν την τομεακή στήριξη δίνονται πρωτίστως Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία, δεν είμαι ιδιαίτερα δημιουργικό, ε, χρησιμοποιώ αυτή που έχουμε στι αναλύσει μα, είναι οι περιοχέ του Νότου. Διότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μια περιφερειακή κατανομή και έτσι χαρακτηρίζονται στι εκθέσει μα. Και ε, δεν σημαίνει αυτό ότι προδικάζω τίποτα όσον αφορά που, την ορολογία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ή που θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα, προσωρινή εφαρμογή. Ο συνάδελφος Φερνάντο μόλις υποθύμησε τη θέση της κυρίας Μάλστρομ για τις εμπορικές συμφωνίες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ελευτικές συμφωνίες σε γενικές γραμμές ε, θέλουμε να έχουμε μια προσωρινή εφαρμογή για να αποφύγουμε το εξή, να διακοπούν οι αλληλευτικές δραστηριότητε ε, των αλέων. Και γνωρίζετε ότι εδώ και κάποια χρόνια υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Και το Κοινοβούλιο, ε, όταν ε, ήταν σε προσωρινή εφαρμογή αυτή η συμφωνία με το Μαρόκο, αποφάσισε να μην ε, δώσει τη συμφωνή γνώμη του, κάτι το οποίο οδήγησε σε κρίση και οδήγησε και σε μήνες αδράνειας για τους αλείς. Τα γνωρίζουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Απ' τη μια υπάρχουν τα συμφέροντα της κάθε πλευράς και θα δράσουμε αναλόγως. Τώρα, όσον αφορά τα γράμματα για την αλληλευτική συμφωνία, όπω σα είπα, οι διαπραγματεύσει έχουν ξεκινήσει. Είμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευση. Σα είπα ότι το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή προβλέπει δραστηριότητε μέχρι τι 14 Ιουλίου ε, τα μεσάνυχτα, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία δραστηριότητα, διότι κανένα σκάφος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα ύδατα ε, της χώρας, εάν δεν υπάρχει συμφωνία και ε, το πρωτόκολλο της συμφωνίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραμπό. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική Δράσης, εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω κι εγώ σε κάποιες ερωτήσεις περισσότερο διπλωματικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα ότι οι διαπραγματεύσεις στι οποίες αναφερόμαστε και που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Ό,τι έχει να κάνει με τη συγκατάθεση και κυρίως τη σχέση μας με το μέτωπο Πολυσάριο είναι περισσότερο πολιτικής φύσεως. Το πολιτικό σκέλος είναι στα χέρια του ΟΕ, για τη Δυτική Σαχάρα. Πάντα αυτή ήταν η στάση μας και παραμένει. Και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε περισσότερο και από ό,τι το κάναμε κατά το παρελθόν τις προσπάθειες του ΟΕ και του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Κέλλερ, για να επιτευχθεί μια ρεαλιστική πολιτική λύση που να είναι αμοιβαία αποδεκτή Υπενθυμίζω ότι το τελευταίο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της ε, εντολής ε, της αποστολής του ΟΗΕ που εγκρίθηκε πρόσφατα αναφέρει όπως και τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια αυτούς τους όρους. Ρεαλιστική πολιτική λύση αμοιβαία αποδεκτή βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή είναι η εντολή του κύριου Κέλλερ. Τώρα, για να επανέλθουμε στην ε, συγκατάθεση και το μέτωπο Πολυσάριο. Το μέτωπο Πολυσάριο είναι ένας ε, σημαντικός ε, συνομολητής στην διαδικασία την ειρνευτική των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζω επίσης ότι το μέτωπο Πολυσάριο δεν είναι απαραίτητο ότι αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τα εμπορικά συμφέροντα των τοπικών πληθυσμών σε μια ουσιαστικά εμπορική διαπραγμάτευση. Είναι ένα σημαντικό εταίρο με τον οποίο έχουμε σχέσεις και επαφές. Για το ποιος έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των, του λαού της Δυτικής Σαχάρας, των πληθυσμών εκεί, Νομίζω ότι αυτό παραμένει ακόμα ανοιχτό ο ζήτημα. Μάλλον δεν υπάρχει τέτοια αποκλειστική εκπροσώπηση. Και ο ίδιος ο ΙΕ δέκα χρόνια, στην αρχή τουλάχιστον των 17 ετών, προσπάθησε να καταφέρει να πετύχει δημοψήφισμα και δεν τα κατάφερε. Δεν είμαστε εμείς σε μια εμπορική διαπραγμάτευση που θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να καταλήξουμε σε έναν και μοναδικό συνομιλητή μας εκεί. Δεν υπάρχει τέτοια αποκλειστική εκπροσώπηση. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το υπενθύμησε στην προηγούμενη απόφασή του, στη γνωμοδότησή του μάλλον, στα πλαίσια της απόφασης για τη Γεωργική Συμφωνία, ότι το μέτωπο Πολυσάριο δεν ήταν σε θέση να εκπροσωπήσει τα εμπορικά συμφέροντα του λαού ή του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, είναι στα χέρια του ΟΗΕ, που στηρίζουμε εμείς και τις προσπάθειές του. Υπενθυμίζω επίσης ότι στην τελευταία απόφαση για την αλληλευτική συμφωνία της 27ης Φεβρουαρίου δεν υπάρχει μνήα του μετόπου Πολυσάριο. Αυτό εξηγεί γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα συνομιλητή, ο οποίος όμως δεν είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων πληθυσμών σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είναι πολιτική. Η πολιτική είναι στα χέρια των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Η συγγήτριά μας τώρα, η κυρία Πατρίσια Λελόντ, θέλει πάλι το λόγο για τις ε, τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα υπόθηκαν εδώ θα προσπαθήσουμε. Κατάλαβα ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην πολιτική και την ε, εμπορική πτυχή. Κάτι το οποίο, εντάξει, είναι το λιγότερο. Αυτή η υπόθεση, εγώ νιώθω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Ακούμε τους συναδέρφους, ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, συμφωνούν οι απόψεις. Ο κύριος Κέλλερ θέλει να μην πληγεί το Μαρόκο στα συμφέροντά του, να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο, αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Όμως, από την άλλη, θέλει η Σαραουή που εκπροσωπούνται από το Πολυσάριο, που ίσως όντως να μην είναι ο μόνος που μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του λαού εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι χάρη στον κύριο Κόλλορ και στο έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή στάση για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση η οποία συμφωνώ ότι, για την, όπως είπε και η Μαρία, είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην έχουμε μια συμφωνία η οποία να καταργηθεί τρεις μήνες αργότερα γιατί δεν θα στέκει. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση και έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 20 έχουμε τα διάφορα. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Όχι. Ωραία. Συνεπώ, δεν έχουμε άλλε σημείε στην ημερήσια διάταξη και έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μα συνεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ όλου. Επόμενη συνεδρίαση. 20 και 21 Ιουνίου εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ.